Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίευα, και καλώς ήρθατε στην ε, συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Ανάπτυξη. Όλοι γνωρίζουμε το στόχο αυτής της συνεδρίασης που είναι η ακρόαση της κυρίας Γεωργίευα για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες της ε, για την ανάλυση των καθηκόντων της Επιτρόπου Αρμόδιας για Διεθνή Συνεργασία, Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων. Το χαρτοφυλάκιο που τη ανατέθηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο. Σας υπενθυμίζω ότι με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 17 του κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί του προτινόμενους επιτρόπους επί τη βάση των γενικών τους ικανοτήτων, της ευρωπαϊκής τους προσήλωσης και δέσμευσης και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Το Κοινοβούλιο επίσης αξιολογεί τι γνώσει του ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό του, καθώ και τι επικοινωνικέ του ικανότητε. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι πριν την ακρόαση η προτινόμενη επίτροπο έστειλε τι απαντήσει τη γραπτό σε ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι γραπτέ απαντήσει έχουν διανεμηθεί. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εν συντομία την διαδικασία αυτής της ακρόασης. Θα ξεκινήσουμε με σύντομες δηλώσεις των πολιτικών ομάδων ως προς τις προτεραιότητές τους ε, σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείριση των κρίσεων. Στη συνέχεια, η προτινόμενη επίτροπος ε, θα προβεί σε μια εισαγωγική δήλωση που δεν θα πρέπει να υπερβεί το δεκάλεπτο Κατόπιν ακολουθούν δύο ώρες και 3 τέταρτα ερωτήσεων ε, ξεκινώντας με ένα γύρο τραπέζης από έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικής ομάδας. Η συζήτηση αυτή θα εκτελεχθεί με βάση την αρχή του πινκ-πονγκ με τρία μισή λεπτά γύρους ερωτήσεων. 45 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση, ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση και μισό λεπτό για συμπληρωματική ερώτηση και 30 δευτερόλεπτα ενδεχομένω για συμπληρωματική απάντηση. Θα ήθελα να σας πεθυμίσω ότι ο χρόνος αγόρευσης των ε, Ευρωβουλευτών περιορίζεται αυστηρά στα 45 δευτερόλεπτα. Όσο πιο σύντομε είναι οι ερωτήσει, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε και τι απαντήσει τη υποψηφία επιτρόπου και ενδεχομένω για υπερωτήσει. Θα ήθελα να σα διευκρινίσω ότι οι συμπληρωματικέ ερωτήσει πρέπει όντω να είναι συναφεί με την απάντηση τη υποψηφία επιτρόπου και δεν θα πρέπει να άπτονται άλλων θεμάτων. Ω πρόεδρο τη Επιτροπή και πρόεδρο τη ε, Συνόδου τη Ακρόαση αυτή, ε, ε, έχω το δικαίωμα να μην δεχθώ συμπληρωματικέ ερωτήσει που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Θα έχουμε λοιπόν δύο σύντομου γύρου ερωτήσεων με βάση το σύστημα Catch the Eye για θέματα που προσδιορίστηκαν από του συντονιστέ και αποτελούν προτεραιότητε τη Επιτροπή μα. Οι ευρωβουλευτέ που θέλουν να λάβουν μέρο στη συζήτηση αυτή θα έχουν μεταξύ 15 και 20 δευτερολέπτων για να θέσουν τι ερωτήσει του και θα ήθελα να θέρμο παρακαλέσω και την υποψήφια Επίτροπο να είναι άκρο συνοπτική απαντήση τη θα δοθεί προτεραιότητα στις συζητήσεις αυτές στα πλήρη μέλη και στα αναπληρωματικά μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μας. Βέβαια προβλέφθηκε και λίγος χρόνος για να μπορέσει η Επίτροπος να διευκρινίσει τις απαντήσεις που έδωσε σε ορισμένες ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών και που δεν έτυχαν ικανοποιητική ή διεξοδική απάντηση. Αυτό θα μας το επισημαίνουν ε, ενδεχομένως οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Επίσης έχουμε προσκαλέσει και τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών Υποθέσεων ε, στην ακρόαση αυτή και θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους μέλη αυτών των δύο επιτροπών. Στο τέλος της ακρόασης θα καλέσω την κυρία Γεωργίευα, την υποψήφια επίτροπο, για μια σύντομη τελική δήλωση, αν το επιθυμεί. Η δερμηνή υπάρχει για όλες τις γλώσσες, οπότε όλοι οι αγορητές μπορούν να μιλούν στη μητρική τους γλώσσα. Σας παρακαλώ όμω δεδομένη της ύπαρξης διερμηνίας, θα ήθελα να επισήσω την προσοχή των Ευρωβουλευτών για να μην μιλούν πολύ γρήγορα. Η ακρόαση αναμεταδίδεται απευθείας στο web stream του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πρακτικά επίσης μπορείτε να τα βρείτε στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκινούμε λοιπόν με τις δηλώσεις των πολιτικών ομάδων, δίνοντας το λόγο πρώτα στον κύριο Κατσμάρεκ για το ΕΛΚ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά θέματα για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Η ανθρωπιστική ενίσχυση αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά με τη συνθήκη της Λισαβόνας ως σημαντική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε επίτροπο που έχει ως ρητή αρμοδιότητα την ανθρωπιστική ενίσχυση. Μάλιστα, η δημιουργία αυτού του χαρτοφυλακίου είναι σημαντικό μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουμε να ενισχυθεί ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα διεθνέ προσκήνιο στα θέματα αυτά. Και αυτό είναι βήμα προ την καλή κατεύθυνση. Είμαστε μεγαλύτερος χορηγό ανθρωπιστική ενίσχυσης ε, στον κόσμο. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον συντονισμό, στη συνοχή και στη συμπληρωματικότητα αυτής τη ανθρωπιστική βοήθειας και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και νέες προκλήσεις που ανακύπτουν στα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Και οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είδαμε την τελευταία θεομηνία, το σεισμό στην Αϊτή. Θέλουμε ε, ουδέτερη και αποτελεσματική χορήγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δυστυχώς ε, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι στα θέματα αυτά, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί, ε, πολλά μέλη προσωπικού στο, στα θέματα τα ανθρωπιστικά χάνουν τη ζωή τους, γιατί είναι εύκολος στόχος. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τέτοια φαινόμενα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπέργκμαν από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κυρία υποψήφια, υποψήφια Επίτροπε, η ανθρωπιστική ενίσχυση, όπως ξέρετε, είναι ένα συνεχής αγώνας μεταξύ της Realpolitik των ισχυρών, με, το με τα στρατηγικά και βιομηχανικά του συμφέροντα, και τις ζωές ε, λιγότερο ισχυρών ε, ανδρών, γυναικών και παιδιών. Οι γυναίκες και τα παιδιά δυστυχώς είναι τα θύματα πρώτης γραμμής στις ε, χώρες αυτές. Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τους πληγέντες, τους αναξιοπαθείς, αυτούς που βρίσκονται ε, σε κίνδυνο ε, έξαρσης μιας νέας σύγκρουσης μόνο και με την άφηξη των ανθρωπιστικών αγαθών ρόλο σα θα είναι να δείξετε αποφασιστικότητα και πυγμή κατά την υλοποίηση των καθηκόντων τη Ένωση. Μερικέ φορέ θα πρέπει να επιβάλλετε το σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου, γιατί πολλέ φορέ ε, δεν είναι προτεραιότητα αυτό για όλου του υπουργού. Μπορεί να ήταν εύκολα τα πράγματα στην ΑΕΤ, να φαίνονται εύκολα, αλλά δυστυχώ ε, οι θεομηνίε δεν είναι πολύ διαφορετικέ από τι ανθρωπογενεί καταστροφέ και το τσουνάμι δεν είναι ταρφούρ. Υπάρχουν πραγματικά διλήμματα και ε, φρικαλαιότητε που ο άνθρωπο επιβάλλει πολλέ φορέ στον ίδιο τον άνθρωπο θα πρέπει να έχουμε τρόπους να επέβουμε και δυστυχώς η μετριοφροσύνη είναι το τελευταίο που περιμένουν από μας τα θύματα και οι πλημμύρες στη Βερμανία δίνουν τα όρια των δυνατοτήτων μας. Η ομάδα μα θα σταθεί στο πλευρό σα για να ενισχύσουμε τι ανθρωπιστικέ αρχέ στον κόσμο, δείχνοντα ότι για την Ευρώπη κάθε άνθρωπο αξίζει ένα αξιοπρεπέ μέλλον. Περιμένουμε λοιπόν τις απόψεις σας για τα πολλά διλήμματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπιστική βοήθεια και θέλουμε επιθυμία να μεταφέρετε από την Ευρώπη μια αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς από τους Φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψηφία Επιτροπέ. Η ανάληψη των καθηκόντων σας ε, συμπίπτει με την απαρχή απάντησης που δίνουμε στην καταστροφή της ΑΕΤΗΣ. Και μάλλον θα είστε η επίτροπος που θα έχετε το λιγότερο χρόνο στη διάθεσή σας για να προετοιμάσετε μία αντίδραση ε, σε ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα όπως είναι αυτό των ανθρωπιστικών θράσεων. Επίσης, ε, οι συνομιλητές σας θα είναι πολύ άριθμοι. 27 χώρες μέλη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχετε τουλάχιστον άλλους δύο επιτρόπους που άμεσα ή έμεσα θα έχουν παρόμοιες δραστηριότητες, οπότε θα πρέπει να συντονιστείτε μαζί τους. Επίσης, υπάρχει και ένα λιγότερο θεαματικό ζήτημα. η μεγαλη ξεχασμενη που είναι οι ασθενείς που περιμένουν ε, μία θεραπεία ε, κατά του ρετροϊού και για αυτούς η δράση σας θα είναι πολύ σημαντική. Τέλος, έχετε απέναντί σας και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιθυμεί διάλογο μαζί σας, προσπαθώντας να εφαρμόσει τη συνθήκη της Λισαβόνας που μας επιβάλλει αυτό το χρέος, το καθήκον συντονισμού σε θέματα ανθρωπιστικών, ανθρωπιστικής βοήθειας και αντίδρασης στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κατρίν Γκρές από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γεωργίευα, η προσήλωσή σας, η δέσμευσή σας, οι ικανότητές σας και οι γραπτές σας απαντήσεις είναι πολύ εθαρρυντικές για την ομάδα μας. Δεν θα σας εκπλήσω ότι μία από τις προτεραιότητες των Πρασίνων είναι η απάντηση που θα δώσουμε στις ε, θεομηνίες που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές. Βέβαια δεν είναι όλες οι θεομηνίες συναφείς με τις κλιματικές αλλαγές όπως έτσι, αλλά η άνοδος του, ε, του επίπεδου του ύδατος, η ανιδρία, η επιτάχυση των ανέμων με κάποια συναφή κλιματολογικά φαινόμενα. Βέβαια η ανθρωπιστική ενίσχυση συνδέεται και με άλλες πολιτικές πρόληψης των κινδύνων που θα πρέπει παράλληλα να εφαρμοστούν. Ερωτώ λοιπόν, ποιες είναι οι συγκεκριμένες σας προτάσεις σε σχέση με την πρόληψη θεομηνιών που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές και πώς θα μπορούσατε να επηρεάσετε τους ε, συναδέλφους σας για να λάβουν υπόψη αυτά τα θέματα. Η ομάδα μας ανησυχεί για την νέα οργάνωση και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και χαρτοφυλακίων για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ το λόγο κύριος Ντέβα από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ήρθατε στην ακρόαση με πλούσια πείρα από τη Παγκόσμια Τράπεζα και αλλού. Η ανησυχητική, η ανθρωπιστική βοήθεια φυσικά είναι απόρρια της ανθρωπιστικής παρέμβασης και η ευθύνη προστασίας είναι από τις σημαντικότερες ευθύνες που φέρουμε ως ανθρώπινα όντα. Παλιά η ευθύνη της προστασίας ε, θεωρούνταν ως επέμβαση στην εθνική κυριαρχία. Πρόσφατα όμως μια τέτοια ευθύνη προστασίας μπορεί να συμβάλλει στην δυνατότητα της ε, εδραίωσης μιας κυριαρχίας και της ε, ενίσχυσης της δυνατότητας που έχει κάθε κράτος να αυτοπροστατευτεί. Πώς θα επέβουμε σε περιοχές όπως τον Ταρφούρ για να ενισχύσουμε το δυναμικό αυτών των χωρών, να αυτό βοηθηθούν. Πώς θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, τις κυβερνήσεις τους, τις αρχές τους για να αναλάβουν την ευθύνη τους, για να κάνουν τα πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν, θα όφιλε να κάνουν, που δεν δίνανται αυτή τη στιγμή. Επίσης, ποιο είναι το μελλοντικό σας όραμα για τις ε, ανθρωπιστικές δράσεις και την ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξέχοντα ρόλο να αναλάβει εδώ γιατί θέλουμε να προσπίσουμε, να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές και να διασώσουμε χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας και να δώσουμε δυνατότητα σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις στον κόσμο να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του για ένα καλύτερο μέλλον. Περιμένουμε λοιπόν τις απόψεις για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει Γκάμπι Τσίμερ από την ΚΟΕ. Um, της αριστεράς. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να αναφέρω τις προσδοκίες μας. ότι η νέα κάλυψη του χαρτοφυλακίου Επιτρόπου για την προστασία από καταστροφές και ανθρωπιστική βοήθεια θα συσχετιστεί γενικά με μια συνεπή πολιτική ανάπτυξης και θέματα που μέχρι στιγμής ήταν εκτός του τομέα αυτού, ιδίως θέματα προληπτικής προστασίας από καταστροφές. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μας παρουσιάσετε τις ηγετικές σας απόψεις. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο βοήθειας προς τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε χώρες που πλήττονται από καταστροφές να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους κάποια ε, κονδύλια που δεν μπορούν να τους δοθούν αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο σκοπεύετε να φροντίσετε να δίνονται επενδύσεις για την δημόσια υποδομή και τις δημόσιες αρχές και κατά πόσον το νέο μέσο για το είδωρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών και να ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο, να διευρυνθεί για να καλύψει και άλλες χώρες, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση χρημάτων για την δημόσια χορήγηση υδάτος. Ευχαριστώ. E Το λόγο έχει ο Μάριο Μποργέζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υποψήφια Επίτροπο στι απαντήσει τη ε, στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την άποψή μου, απέφυγε να απαντήσει σε μια από τις ερωτήσεις που ήταν λογικό να περιμένουμε να απαντήσει με την ευκαιρία αυτή της ακροασίας. Πώς κρίνεται την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά τις μέρες αμέσως και τις εβδομάδες που ακολούθησαν την τραγωδία της ε, IT που για πολλές μέρες και ίσως και κάποιες εβδομάδες αποτέλεσε το μαύρη τρύπα του, της υφηλίου και προσέφερε δυστυχώς ένα αρνητικό θέαμα μαζικών παρεμβάσεων που ήταν όμως ασυντόνιστες. Όλα αυτά κόστησαν πολύ στις χώρες και στις κυβερνήσεις αλλά σίγουρα δεν έδωσαν τα αποτελέσματα που περιμέναμε και που θα μπορούσαν να έχουν. Διερωτώ με, τι χρησιμεύουν όλα αυτά τα πακέτα βοήθειας που πετιούνται από ψηλά χωρίς καμιά λογική. Ίσως ε, θα έπρεπε να, δοθούν, ε, να βοηθούν μάλλον ε, τους πιο οπλισμένους, τους πιο ισχυρούς, αλλά σίγουρα όχι τους, αυτούς που χρειάζονται τη βοήθεια. Επίσης, τι μπορείτε ακόμα να μας πείτε για ορισμένα θέματα. Θεωρείτε πως είναι απαραίτητη μια μεγαλύτερη διαφάνεια στο ποιος ενεργεί συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, γιατί στην ΑΕΤ βασικά ασχολήθηκαν με το να προβάλλουν ε, τα σήματά τους στις τηλεοράσεις σε ολόκληρο του κόσμου και ε, κλείνω με το ρόλο της στρατιωτικής παρέμβασης σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Πρόεδρος, ο λόγο έχει τώρα η υποψήφια Επίτροπος για τη δήλωσή της, την ε, εισήγησή της για 10 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε μόνιμε εισηγητή, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, είναι τιμή μου και προνόμιό μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ ως υποψήφια επίτροπος για την διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων. Είναι επίσης μεγάλη ευθύνη για αυτούς που περισσότερο έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο της Κομισιόν. Με τη δημιουργία του η Ένωσή μας αναγνωρίζει μία ατυχή τάση, την ε, Ε, αύξηση το, της συχνότητας και της έντασης των φυσικών και ανθρωπογενών ε, καταστροφών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνδυαστεί η ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και η ανταπόκριση της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να συμβαδίζουν και ε, μια μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από το 90% των πολιτών μας θέλουν να δουν την Ευρώπη να επιταχύνει και να βελτιώνει ε, τις προσπάθειές της για ανταπόκριση και ενίσχυση σε φυσικές ε, καταστροφές ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα βρισκόμαστε στα μέσα μιας κρίσης που κόστησε τη ζωή σε πάνω από 150.000 αιτινούς. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την οδύνη και την οδύνη όλων αυτών που επλήγησαν και τη δική μας για εκείνους. Πριν από το σεισμό τον Ιανουάριο, στις 12 Ιανουαρίου η ΑΕΤ ούτως ή άλλως πάσχει να ξεπεράσει την, το κληροδότημα διαφθορτικών προβλημάτων και τον αντίκτυπο των τυφών 2008. Η ΑΕΤ ξεκινά από το μηδέν, αλλά δεν είναι μόνη. Εάν με επικυρώσετε θα είναι άμεσό μου καθήκον να διασφαλίσω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα προσφέρουμε στην ΑΕΤ ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η Ένωσή μας. Μάλιστα, εξέτασα την ανταπόκριση της Κομισιόν και των κρατών μελών και με εντυπωσίασε το έργο των ανθρώπων μας επιτόπου η ανθρωπιστική μας βοήθεια και οι υπηρεσίες της μαζί με τις υπηρεσίες ε, της ε, προστασίας των πολιτών ενέργησαν άμεσα. Η Κομισιόν απελευθέρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ και το προσωπικό μας ήταν επιτόπου. Τη δεύτερη μέρα οι δικοί μας εκπρόσωποι διαβεβαίωσαν ότι δεκάδες χιλιάδες αιτινοί είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 25 ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν ε, την στήριξη που χρειαζόταν μέσω του, κέντρου συντονισμού και βέβαια τις πρώτες μέρες αυτός ο συντονισμός δεδομένου ότι ο ΙΕ με πολύ πραγματικό και τρόπο βρισκόταν στην ΑΕΤ και δυστυχώς ο υπεύθυνο του ΙΕ έχασε τη ζωή του, οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες. Όπως πάντοτε η Ευρώπη έδειξε Μεγάλη γενεοδορία δέσμευσε 500 εκατομμύρια για να, την άμεση ανακούφιση και τη βοήθεια για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι ένας εντυπωσιακό αριθμός ιδιωτικών δωρεών έδειξε την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων πολιτών με αυτούς που την χρειάζονται. Υπάρχουν τώρα δύο έργα προτεραιότητα στην ΑΕΤ. Καταρχήν να ενεργήσουμε αποφασιστικά και να, δώσουμε, να συνεχίσουμε να δίνουμε άμεση ε, βοήθεια, ιδιαίτερα στέγη, τροφή και υπηρεσίες υγειονομικές και δεύτερον να ξεκινήσουμε τη δουλειά στο να να, να ενσωματώσουμε την ε, βοήθεια με την ανοικοδόμηση. Όλα αυτά ξέρουμε πως θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η κυβέρνηση της ΑΕΤ θα μπορέσει να αναλάβει και να παίξει ηγετικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο κινητοποιούμε 100 εκατομμύρια ευρώ για μη ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίω για να βοηθήσουμε να αποκατασταθούν οι λειτουργίε τη κυβέρνηση και οι υπηρεσίε τη. Την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν θα συμμετάσχει σε μια διεθνή αποστολή προς, στην ΑΕΤ για να προετοιμαστεί μια ε, κοινή εκτίμηση αναγκών, πράγμα που θα κατευθύνει τις συλλογικές μας προσπάθειες για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, μετά τη Χαϊτή, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα που είναι στο μυαλό όλων και το έχουμε ακούσει αυτό το ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για ταχύτερη, πιο ενωμένη, πιο ορατή Ευρώπη όταν θα χτυπήσει η επόμενη θεομηνία. Εγώ με μεγάλη χαρά είδα ότι την επόμενη εβδομάδα οι ικανότητες ανταπόκρισης της κρίσης της Ένωσης θα είναι στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εγώ δεσμεύομαι πως θα, συνεχίσω, θα παρακολουθήσω μάλλον τις συζητήσεις του Συμβουλίου ενεργά και θα ζητήσω κατευθύνσεις και από την έκθεση Μπαρνιέ του 2006 που μάλιστα έχει γίνει έχει αποτελέσει το γνώμονα για πολλές ενέργειες, αλλά δεν έχουμε ακολουθήσει όλες τις λεπτομέρειες. Και βεβαίως ε, θα ήθελα να αναζητήσω μια ευκαιρία να συζητήσω τα θέματα αυτά με την Επιτροπή σας όσο γίνεται πιο σύντομα. Φυσικά αν με εγκρίνετε. Κύριοι βουλευτές, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που μοιάζουν με την ΑΕΤ, όπου ένας ε, τυφώνας, μια πλημμύρα ή μια σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ζωών και να οδηγήσει εκατομμύρια ιδιαίτερα γυναίκε και παιδιά στην ε, άκρα παινία. Είτε είναι μαζικές πλημμύρες στο Μπαγκλαντές, είτε είναι η σύγκρουση στο Σουδάν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο κόσμος είναι που υποφέρει. 300 εκατομμύρια ετησίως επηρεάζονται από φυσικές δομηνίες ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Είναι εντυπωσιακό ο αριθμός. 42 εκατομμύρια τουλάχιστον άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο εντός της χώρας τους ή εκτός. Και αυτοί οι αριθμοί θα αυξηθούν λόγω των κλιματικών αλλαγών, λόγω της ταχείας αστικοποίησης και λόγω της, ε, του χαρακτήρα πολλών κρατών. Αυτές είναι οι υποσχέσεις που εγώ μπορώ να σας δώσω σήμερα, αν με εγκρίνετε. Θα προσπαθήσω να έχω ισχυρή φωνή ε, υπέρ των όσων ε, ε, έχουν ανάγκη. Θα προωθήσω τις προτεραιότητες που έχουμε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, πιο αποτελεσματική βοήθεια, καλύτερες δυνατότητες ανταπόκρισης, βελτιωμένος συντονισμός εντός της Ένωσης και ανάμεσα στους ανθρωπιστικούς και τους στρατιωτικούς φορείς, που είναι πολύ περίπλοκο ζήτημα, αλλά πολύ σημαντικό θα σταθώ υπέρμαχος του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και επίσης θα ορθώσω το ανάστημά μου όταν σκοτώνονται εργαζόμενοι των ανθρωπιστικών ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας όταν ε, γίνεται κατάχρηση των ε, κρατουμένων και όταν χρησιμοποιείται σεξουαλική βία ως όπλο, πολεμικό όπλο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποδώσω στην δέσμευσή μας να περιοριστούν οι κίνδυνοι θεομηνιών καθώς και θα αναθεωρήσω και θα ενισχύσω το μέσο για την προστασία των πληθυσμών. Θα εφαρμόσω την εντολή της συνθήκης της Λισαβόνας για, παροχή, για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών ανθρωπιστικών, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και θα προσφέρουμε και ένα σύνολο εμπειρογνωμοσύνης για τις ανθρωπιστικές μας προσπάθειες καθώς και μια βάση που θα συγκεντρώνει τις δικές μας ευρωπαϊκές αξίες. Και τέλος ε, θα ενεργήσουμε έτσι μαζί με το σύνολο των επιτρόπων ώστε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας πιο αποτελεσματικά και οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι περήφανοι για την ε, ανθρωπιστική ε, βοήθεια και την ανταπόκριση στις κρίσεις. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή όπου αυξάνονται οι ανάγκες και υπάρχει πιο έντονος ανταγωνισμός για πως εντό τη Ένωση για ολόκληρη την ατζέντα της ανάπτυξης. Όλα αυτά καθιστούν το έργο της Κομισιόν και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και με τους άλλους εταίρους πολύ σημαντικά. Εντό τη Κομισιόν με στενή συνεργασία με την Βαρόνη Άστον και τον κύριο Πίμπαλ θα μου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσω το πλήρες δυναμικό ε, της Κομισιόν για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Επίσης θα συνεργαστώ με τους τους ε, υπόλοιπους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τις εσωτερικές υποθέσεις, το περιβάλλον, τις ε, ενέργειες για το κλίμα και στον τομέα της ανταπόκρισης της κρίσης. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, η μακρά μου εμπειρία στην ανάπτυξη, στην αναπτυξιακή βοήθεια, μου έχει δώσει το εξή δίδαγμα. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Όμω, ε, με συνεργαζόμενοι μπορούμε να σημάνουμε τη διαφορά. Και με αυτή την ε, πεποίθηση προσεγγίζω τη σημερινή ακρόαση και αν με εγκρίνετε θα επανέλθω στην Επιτροπή σας ώστε να με κατευθύνετε και στο μέλλον. Και οι ερωτήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες. Ευχαριστώ. Nous avons maintenant notre première θα περάσουμε τώρα στον το γύρο Catch the που έχει σαν θέμα το ανθρωπιστικό έλλειμμα, ανθρωπιστικό κενό. Δηλαδή η απαραίτητη ανάγκη συντονισμού των διαφόρων και στο ιστορικό τη Κομισιόν, ανθρωπιστική βοήθεια, ανάπτυξη και άλλοι παράγοντε εξωτερικής μας δράσης. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης. Ερωτήσεις παρακαλώ. Το λόγο έχει ο κύριος Εξέλ. Ευχαριστούμε κυρία Γεωργίευα. Ένα σημαντικό τμήμα των Σαχαροϊτών ε, χρειάστηκε να εκπατριστεί, βρίσκεται σε καταβλισμούς ή στην Αλγερία ε, θα κάνετε κάτι προκειμένου να προσφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς τους αχαραοίτες που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους. Η υποψήφια Επίτροπος έχει το λόγο. Στην ε, Κομισιόν, στην Γενική Διασέκο, έχουμε φροντίσει να μην ξεχνάμε τις κρίσεις ε, που έχουν διαρκέσει τόσο πολύ. Αναφερόμαστε εδώ σε πληθυσμό που υποφέρει για μακρά χρονικά διαστήματα λόγω δυσκόλων οικολογικών συνήθω ε, προποθέσεων. Το πιο σημαντικό είναι να μην του ξεχάσουμε. Πάντα να τους έχουμε κατά νου, πάντα να γνωρίζουμε τι ανάγκε τους και οπωσδήποτε αυτό θα είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα μου. Και αυτό που κάνουμε είναι να έχουμε ένα κονδύλι για τις λεγόμενες ε, ξεχασμένες κρίσεις. Είναι κάτι που είναι σημαντικό κατά μένα και θα θέλω να το συνεχίσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. In Sudan, the first recipient of... Η πρώτη που έλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν, κύριε ήταν εκείνη που παρατηρούσαν τις εκλογές όπου ο κ. Αντεσίρ θα πρώτη να εκλεγεί στην Αιθιοπία πάλι μια μεγάλη χώρα υποδοχής ε, ενίσχυας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί και τις εξωγές όπου υπάρχουν προβλήματα. Η πρόεδρος διακόπτη. Πώς θα φροντίσετε να υπάρχει μια συνοχή, συνοχίζει ομιλήτρια χωρίς μικροφόνου. Δεν έχετε το λόγο. Η κυρία Επίτροπος, μήπως μπορείς να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Το επίκεντρο της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η ουδετερότητα και η φροντίδα για τους ανθρώπους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι εκείνοι που υποφέρουν χωρίς να έχουν ασφάλει ήδη συχνά να λάβουν βοήθεια. Και έχουμε διάφορα μέσα για να μπορέσουμε να ασχίσουμε πίεση στις κυβερνήσεις. Στην περίπτωση του Σουδάν, όπως ξέρουν όλοι νομίζω εδώ οι παρόντες, δεν υπάρχει καμία αναπτυστική βοήθεια. Δεν έχουμε συμφωνία. Ε, δεν έχουμε συμφωνία κοντονού μαζί τους για καλούς λόγους ή να πούμε για κακούς λόγους. Να προσπαθούμε να βοηθήσουμε ε, θύματα πολέμων ή, ή φυσικών θεομηνιών. Πάνε η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι βοηθησουμε θυματα πολεμων η η όσον αφορά την πολιτική διάσταση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η ανθρωπική βοήθεια να βρεθεί στα χέρια εκείνων που καταχρώνται της εξουσίας. Και γι' αυτό εργαζόμαστε με τις ε, ε, οργανώσεις επιτόπου και όχι με τις κυβερνήσεις. Η κυρία Κριτού έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που μου είπατε με διέφεραν πάρα πολλά γιατί Αναφέρατε συγκεκριμένα την κατάσταση στην ΑΕΤ, γιατί ακριβώ η δική σα εντολή θα αρχίσει με την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση της αντιμετώπισης αυτής της έκτακτης ε, συγκυρία σε αυτή τη χώρα. Και η ερώτησή μου είναι η εξή πώ θα περιγράψετε την αποτελεσματικότητα μεταξύ βοήθεια και ανάπτυξη και πώ θα συνεργαστείτε με τον Επίτροπο για εξωτερικέ υποθέσει και τον Επίτροπο για την Ανάπτυξη. Η υποψήφια επίτροπο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Χθες ε, για πρώτη φορά συνάντησα, με το, συνάντησα την υποψήφιο επίτροπο για την ανάπτυξη και ακριβώς αυτό το θέμα συζητήσαμε. Πώς θα φροντίσουμε στην ΑΕΤ να συνεργαστούμε με συνοχή στενά. προβλέπουμε οι ανθρωπιστικές ανάγκες θα παραταθούν. Δηλαδή θα, θα υπάρχει πολλής χρόνος στον οποίο θα χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια και εμείς χρειαζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε επίσης τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης. Πάντα έχουμε αυτό το δίλημα. Την επιλογή δηλαδή μεταξύ ε, βιωσιμότητας και ταχύτητας. Για να βοηθήσουμε του ανθρώπους πρέπει να είμαστε γλίγοροι. Για να διατηρήσουμε όλε αυτέ τις προσπάθειε πρέπει να συνεργαστούμε με τι κυβερνητικέ αρχές. Και ξέρουμε ότι οι κυβερνήτικέ αρχέ στην ΑΕΤ επλήγησαν εξίσου όπω και το υπόλοιπο τη χώρα. Διαβλέπω λοιπόν εδώ ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα από την συνοχή που εδόθη στην κατάσταση του τσουνάμι. Με συγχωρείτε κύριε Γεωργίβα. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο. Climate change is a phenomenon we, we produced, the developed world, but it's affecting the most the Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, η πυρκαγιέ προέρχονται από εμά, αλλά είναι θέμα που πλήγει τι ανεπιστόμενε χώρε. Αυτό οδηγεί εν μέση μέρη και σε ένδια στην προγραμματική κλπ. Γνωρίζετε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν σχετικά για την αναδάσωση και την αντιμετώπιση αποσύλωσης. Υποψήφια Σα ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλή το θέμα αυτό. Μέσα όταν ήμουν στην ε, ε, Διεθνή Τράπεζα σαν Διευθύντρια για το Περιβάλλον προσπάθησα να εξτάσω το θέμα αυτό, την αποφυγή της αποψήλωσης, γιατί πιστεύω ότι αν χάσουμε 20% των δασών, τα προβλήματα ε, στη σχέση με το περιβάλλον είναι τεράστια και θα πρέπει να βρούμε άλλη τόση λύση. Αυτό δεν είναι όμως τη δική μου ε, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, είναι στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου που θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη. Γιατί ξέρουμε ότι η μείωση των δασών μειώνουν την αγροτική α, εξέλιξη και αυτό οδηγεί σε διαμάχες και γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά σε ευρία είναι να τεθεί το θέμα της οικολογικής αηφορίας, αλλά συγκεκριμένα το θέμα της αποψήλωσης και την υποστήριξη της αναδάθωσης. Θα πρέπει να είναι σημαντικό τμήμα της ε, ανάπτυξής μας. Ε, σας ζητώ συγγνώμη που προηγουμένως ε, ξεπέρασε το χρόνο. Η κυρία Βέρστε Γιούγκ, τελευταία ερώτηση αυτής της, αυτού του γύρου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να Είμαι ε, ε, σίγουρη ότι έχουμε μια συντονισμένη και συνεπή πολιτική για την ανάπτυξη εδώ. Για τι συμφωνίε αλληλεία και εμπορίου επίση, γιατί και εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση της ανάπτυξη. Η υποψήφια επίτροπο για το λόγο. Πάλι, αυτό δεν είναι ένα θέμα που είναι του δικού μου χαρτοφυλακίου, δεν θα είναι δική μου ευθύνη, αλλά χάρηκα πολύ που ο πρόεδρος Παρόσο καλεί όλους τους επιτρόπους να συνεργαστούν, να είναι μια ενότητα και οπωσδήποτε θα προωθήσω αυτή την διάσταση, αυτή την πτυχή, να σχεστεί δηλαδή η ένδια που οδήγεται σε περιβαλλοντολογικέ καταστροφές με τη δική μας ανθρωπιστική βοήθεια και οτιδήποτε άλλο κάνουμε να μπορεί να συσχετιστεί με την εντόση αυτών των προβλημάτων. Πάλι δεν είναι δική μου άμεση ευθύνη, αλλά στο Κολέγιο των Επιτρόπων από κοινού θα συνεργαστούμε σαν μία ομάδα. Και θα, υπο, θα χρησιμοποιήσω εκεί την πίθο μου, την επαγγελματική μου εμπειρία σε σχέση με το δικό μου χαρτοφυλάκιο βέβαια. Ευχαριστώ. Πρώτα, θα αρχίσουμε τώρα τον πρώτο γύρο απαντήσεων. 45 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για τις απαντήσεις. Ο κ. Καμιτσάκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να χαιρετήσω τον υποψήφιο ε, επίτροπο. Θα σας πω ε, γιατί είναι περήφανη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες μας είναι ο πρώτος μεγαλύτερος δωρητής ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά δεν φαίνεται έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τους Αμερικανούς αφενός και μετά λέμε τους Γάλλους, τους Γερμανούς, δεν ξέρω. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση ούτω ώστε σε μια περίπτωση χαϊτής να μπορεί ο πολίτης της Ευρώπης να είναι περήφανος, να βλέπει τη σημεία του εκεί ως Ένωση. Τι θα κάνετε για να προοπτευτεί κάτι τέτοιο. Κατερχήν, θα ήθελα να σας πω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να είναι περήφανοι για το τι κάνουν γιατί το 60% της αναπτυσσιακής βοήθειας δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 50% από την ανθρωπιστική βοήθεια. Πέρα από αυτό, η Ευρωπαίοι δίνει κάποιες δυνατότητες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας. Αν εξετάσετε την έκθεση Μπαρνιέ, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν πολύ καλές ε, προτάσεις για να τη βελτίωση του συντονισμού. Και η ερώτηση που υπέβαλα στους ελπίζω μελλοντικούς μου συναδέρφους ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Ε, αυτό δεν θέλετε στο γεγονό ότι οι ορισμένε χώρε έχουν διαφορετικέ προοπτικέ στο θέμα αυτό. Υπάρχει και η αρχή τη επικουρικότητα που λέει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε στο επίπεδο τη Κομισιόν κάτι που θα μπορούν να κάνουν χώρε στο δικό του επίπεδο. Τούτο λεχθέντο και γνωρίζοντα όσο γνωρίζουμε <clears throat> ότι αυτές ε, ε, οι πλημμύρε παραδείγματο του αιώνα θα είναι πολύ πιο συχνά πια από ότι μία φορά σε έναν αιώνα, θα πρέπει να έχουμε μία πιο συνεπή, πιο ολοκληρωμένη, πιο δομημένη θα έλεγα βοήθεια. Συγκεντρωμένη θα έλεγα, όχι όχι, ε, διαρθρωμένη προσέγγιση για να δούμε πού υπάρχουν τα κενά και να τις ενώσουμε. Και μετά βέβαια θα ήταν πάρα πολύ ωραίο εάν εμείς είμαστε Ευρωπαίοι και Βούλγαροι. Για μας τους Βούλγαρους είναι πολύ εύκολο. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, μας αρέσει πάρα πολύ η Ευρώπη, παντού βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε την ευρωπαϊκή σημαία, αλλά χρειάζεται πάλι να συνεργαστούμε για να πείσουμε τις χώρες ότι αυτό έχει νόημα. Ένα και δεύτερο να κατανοήσουμε τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να συνενώσουμε καλύτερα τις χώρες και να προχωρήσουμε σαν μία ενωμένη ενότητα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Βλέπω, πάλι ξεπέρασα το χρώμα μου. πραγματική ερώτηση, κύριε Σμίτσελ. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Ξέρετε ότι έχουμε διάφορες προτάσεις για διάφορες ομάδες ε, διάφορες ε, μονάδες ε, στρατιωτικές, γιατί να μην έχουμε κάτι και στον τομέα αυτό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Για να δουν πραγματικοί οι πολίτες της Ευρώπης ότι με τα λεφτά που πληρώνουν καταφέρνουν πολλά πράγματα απάντηση. Αυτού του τύπου ερώτηση ε, με κάνει να πω ότι είναι καλό να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της ε, Βαρόνης Άστρων, των άλλων υποτρόφων και εμού, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανθρωπιτική βοήθεια. <clears throat> γιατί το θέμα της στρατιωτικής παρέμβασης είναι μια λύση τελευταίας, ε, τελευταίας βαθμίδας, αν θέλετε και θα είναι καλό να χρησιμοποιούμε δυνατότητες που δεν υπάρχουν διαφορετικά. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπέρμαν έχει μια ερώτηση. Κύριε Υποψήφια Πρόεδρε, ε, Επίτροπε, η κατανομή των χαρτοφυλακίων στις εξωτερικές σχέσεις θα καταστήσει δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάμε μία φωνή, όπως ήταν ο στόχος της Συνθήκης Λισαβόνας. Δηλαδή, αναπτυξιακή βοήθεια στα χέρια της ε, κυρίας Άστον, το Ταμείο Ανάπτυξης στα χέρια του κυρίου Μπίμπακ. Υπάρχει συνέπεια. Εκεί πίσω ο κύριος Μπαρόζο να αλλάξει τα πράγματα, να δώσει και τα δύο μέσα αυτά σε έναν ε, και να δώσει ένα ρόλο υποπτία στην είπα το εκπρόσωπο. Εσείς πώς βλέπετε το δικό σας ρόλο ανάμεσα στους δύο συναδέλφους σας. Εγώ θεωρώ ότι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο υπάρχει μεγάλο ποσοστό εσωτερικής λογικής. Καταρχήν δίνει μια φωνή στους άφωνους. Δηλαδή τον υπάρχω εγώ εκεί είναι προς όφελος εκείνων τους οποίους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Δεύτερον, είναι λογικό χαρτοφυλάκιο γιατί είναι ε, ομοιόμορφο ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία των πολιτών. Ταιριάζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα δύο. Και όταν σκέφτομαι την ε, διεθνή συνεργασία, το σκέφτομαι σαν κάποιον ο οποίος είναι υπέρμαχος της ανθρωπικής βοήθειας. Όχι ανθρωπιστική διεθνή συνεργασία, έτσι γενικά και όριστα, αλλά τι μπορεί να γίνει για να βοηθήσουμε συγκεκριμένα προς περιοχές όπως η Ασία, η Λατινική Αμερική που υπάρχουν πολλές φυσικέ καταστροφές ή ε, περιφερειακές ε, οργανώσει όπως η ΑΖΕΑΝ, πόσο χρήσιμο ήταν αυτό στην περίπτωση της Βερμανίας, ε, παραδείγματος κάνει μια επαφή με την Αραβική Λίγα. Εγώ εκεί έτσι βλέπω τον εαυτό μου. Όσον αφορά την οργάνωση του υπολείπου του χαρτοφυλαίου, να σας πω, εγώ προέρχομαι από μια οργάνωση που τα τελευταία ε, δέκα χρόνια ζούσε μέσα σε μια κλίμακα. Δηλαδή οι συλλογικές απαντήσεις είναι κάτι ε, που είναι γνωστό τούτο λεχθέντος πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι τα τετραγωνάκια στα οποία έχει ενταχθεί ο καθένας αλλά η δέσμευση εκείνων που βρίσκονται εκεί να πετύχουν κάτι περισσότερο. Και έτσι πραγματικά είχα την εντύπωση και η Βερόνια Άστον χθε ήταν πάρα πολύ ανοιχτή για να πετευχθεί μια συνεπής προσέγγιση. Και πιστεύω ότι αυτό θα το πετύχουμε πραγματικά. Συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Μπέρκμαν. Σίγουρα θα είναι επικοδομητική συμβολή τη κυρία Άστον και θα δώσει φωνή σε αυτού που δεν έχουν φωνή. Αυτό είναι και ένα σύνθημα που το χρησιμοποιήσω και εγώ γιατί δούλεψα στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια. Να δώσουμε φωνή σε αυτού που δεν έχουν φωνή. Πολύ σπάνια όμω ανθρωπιστικοί διάδρομοι εφαρμόζονται. Το ξέρετε αυτό από την εμπειρία σα στην Ηνωμένα Έθνη τι μπορείτε να κάνετε για να φέρετε ανθρωπιστική ανακούφιση σε έφραυστες περιοχές όπως είναι η Σομαλία. Θα πρέπει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τον εαυτό τη τι γίνεται με την εντολή του ΟΗΕ. Ποιο είναι το δίλημα που αντιμετωπίζετε. Η υποψήφια επίτροπος. Όντως δύσκολη αυτή η ερώτηση. Γιατί όταν συμπεριλαμβάνεται και το στρατιωτικό σχέλος είναι σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και το προσωπικό το, της ανθρωπιστικής βοήθειας λέει το στρατιωτικό να είναι μόνο το τελευταίο καταφύγιο, η ίστατη ε, ενίσχυση. Και στη Σομαλία ανακύπτει αυτό το δίλημα. Εγώ προτιμώ, χρησιμοποιώντας αυτή τη γέφυρα που προσφέρει η κυρία Άστον στους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, να φέρουμε σε αυτή τη χέφυρα και την φωνή από την κοινότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν λέω ότι δεν έχουν φωνή, γιατί είναι ισχυροί άνθρωποι και μιλούμε για τον εαυτό τους, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο. Ο κύριος Γκέρενς. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ήδη στην εισαγωγική σας ομιλία δεχθήκατε την αρχή μιας επιχειρησιακής διάστασης ε, της πολιτικής και ανθρωπιστικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ερώτησή μου αφορά την ε, σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού. Ένας οργανισμός ε, μπορεί να στηρίζεται στις συνεισφορές των κρατών μελών. Πώς θα φροντίσετε να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν χρήσιμα τα κράτη-μέλη στον οργανισμό αυτό, ώστε να ενισχυθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα μπορούσαμε να το είχαμε αξιοποιήσει και στην ΑΕΤ, αν υπήρχε τέτοιος οργανισμός προηγουμένως. Η υποψήφια Επιτρόπος. Έχω την αίσθηση ότι ο, ο μηχανισμός ε, συντονισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσω των κέντρων παρακολούθησης των πληροφοριών επιτελεί στο έπακρο το έργο του, γιατί το έργο του είναι ο συντονισμός και όταν λαμβάνει η χώρα μια θεομηνία μεταδίδονται οι πληροφορίες στα κράτη-μέλη αμέσως και γίνεται μια απογραφή των αναγκών στα κράτη-μέλη να μην στέλνουν ότι ε, έχουν, αλλά ότι χρειάζεται πραγματικά. Φυσικά χρειαζόμαστε μια πιο συγκροτημένη προσέγγιση και φυσικά χρειαζόμαστε και τη συνεισφορά των κρατών μελών. Και η πείρα μου έχει διδάξει ότι μερικέ χώρε είναι υπέρ αναφανδών μια τέτοια πρόταση, άλλε χώρε έχουν επιφυλάξει και οι υπόλοιποι δεν έχουν γνώμη. Και στην περίπτωση της ΑΕΤ εντατικοποιήθηκε η συζήτηση σχετικά. Βέβαια, εγώ ε, αισθάνομαι την ευθύνη να εγκύψω στο θέμα αυτό πιο αντικειμενικά και να δούμε τα υπέρ και τα κατά μιας τέτοιας πρότασης και να προωθήσουμε τη συζήτηση. Και η ιδέα αυτή νομίζω υπευλήθη το 2003 για το EU Fast. Βρισκόμαστε ήδη στο 2010. έχει για κάποιο λόγο μάλλον δεν έχει προωθηθεί νωρίτερα αυτό το σχέδιο. Νομίζω ότι θα ήταν λαζονικό και υπεροπτικό από πλευρά μου να αναπτύξω περισσότερο αυτό το θέμα. Συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Γκέρεν. Πιο συγκεκριμένα. Θα εμπνευστείτε από τη μέθοδο που ήδη ίσχυσε και ήταν αποτελεσματική στην εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας, προκειμένου να γίνει ένα κατάλογο των ικανοτήτων που χρειάζεται για να παρέμβει κανεί σε μια δεδομένη κατάσταση. Δηλαδή, κάθε ε, κράτος να προαναγγέλει τη συμβολή του ανάλογα με τα, τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον κατάλογο αυτό. Η υποψήφια επίτροπος. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η προσέγγιση. Αν γίνει μια χαρτογράφηση των υπαρχουσών ικανοτήτων και τότε μόνο να δούμε τι για να υπάρχουν, δεδομένη και τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο το καλύτερο. Το θέμα είναι αν ο καθένα χρειάζεται ταυτόχρονα να αξιοποιήσει για τον εαυτό του αυτέ τι ικανότητε που έχει. Και δεν μπορεί να συνδράμει άλλου. Τότε είναι που θα πρέπει να επισέλθουμε σε πιο εμβριθή συζήτηση. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Κυρία Γεωργίεβα είπατε ότι δεν μας ενδιαφέρουν εδώ τα κουτάκια, αλλά ο συντονισμός και ο στόχος. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν και ένα σκέλος θα το αναφέρω κι εγώ. Ε, είστε υπεύθυνοι και για την διεθνή συνεργασία, όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τι σημαίνει διεθνή συνεργασία, ποιες είναι οι ευθύνες σας, οι αρμοδιότητες σας εκεί. Η ανάπτυξη, η ανακούφιση, ανασυγκρότηση, ανοικοδόμηση. Γιατί εσείς βλέπετε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συμφωνώ. Το θέμα είναι ποιος είναι αρμόδιος, γιατί ακριβώς. Και τι και εγώ ως Ευρωβουλευτής ήθελα να διαχωρίσουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Η υποψήφια επίτροπος. Η προσέγγιση μου είναι εξή και το συζήτησε και με τη Βαρόνια Άστον και φαίνεται ότι συμφωνεί. Την κρίνει η λογική αυτή την προσέγγιση. Ο ρόλος μου στη διεθνή συνεργασία αφορά πρώτα απ' όλα την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, αντιμετώπιση των κρίσεων, των θεομηνιών. Αυτό είναι το επίκεντρο των αρμοδιότητων μου. Ανακούφιση και παροχή συνδρομής. Και να χρησιμοποιήσουμε ένα απτό παράδειγμα. Όταν είχαμε δυσκολίες με την παροχή βοήθειας στη Βερμανία, στο λαό της Βερμανίας, εκεί τότε έγινε η συζήτηση να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στρατιωτική δράση. Τότε είχαμε διαβήματα προς την ΑΣΕΑΝ, συζήτηση με την ΑΣΕΑΝ και η ΑΣΕΑΝ βοήθησε το προσωπικό, το ανθρωπιστικό, να φτάσει επί τόπου και να βοηθήσει τον κόσμο. Αυτή είναι και η δική μου ιδέα να υπάρξει μια πιο δραστήρια διεθνής προσέγγιση της συνεργασίας και να δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν εταιρικέ σχέσεις για να διευκολύνουμε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των θεομηνιών. Αναφυσβήτητα, αυτό που θα έχουμε στο μέλλον δυστυχώς θα είναι όλο και περισσότερες ανάγκες να αντιμετωπίσουμε θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Πώς θα ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας στα θέματα αυτά. Οχ, εξαντλείται και ο χρόνος μου. Όταν ο Αγγέλαδος χτύπησε την Αιτή, μάλλον όταν ε, χτύπησε το τσουνάμι, το παλιριακό κύμα, αυτό δεν έγινε αμέσως. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα και αν είχαμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα είχαμε σώσει πολλές ζωές. Θέλουμε μια δραστήρια προσέγγιση της διεθνούς συνεργασίας. Και αυτό το σκέλος θα αναπτύξω στις δικές μου αρμοδιότητες. Συμπληρωματική ερώτηση της κυρίας Αργεντίνη δεν θα εξαντλήσω τη δυνατότητα αυτή γιατί έχουμε υπερβεί το χρονικό μας όριο δυστυχώς και και η ερώτηση και η απάντηση. Η κυρία Έμα Μαρκλάρκιν από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το έργο τους. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία προαιρετικής αδειοδότησης και να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ή όχι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έτσι ενισχύεται η διαφάνεια και ο ελεκτικό ρόλος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα βελτιωθεί και η ποιότητα των υπηρεσιών των ΜΚΑΟ. Ποια είναι η δική σας γνώμη για την ε, αντιμετώπιση των ΜΚΑΟ. Στο θέμα της ανθρωπιστικής ενίσχυσης, όλο το έργο δρομολογείται μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Νομίζω ότι έχουμε 186 εταίρους μη κυβερνητικές οργανώσεις που ελέγχονται και αποδεικνύουν τα προσόντα τους ε, για να γίνουν εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Πριν από λίγο ακούσαμε μία ερώτηση για την ευθύνη, για την απόδοση ευθυνών και τη λογοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ένα πολύ σοβαρό σύστημα περιοδικών ελέγχων και επιθεώρησης. Παρακολουθούμε τους εταίρους μας και τα προγράμματά τους, ώστε να να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είτε στον έλεγχο παρουσιάζουν αδυναμίες, είτε τα προγράμματά τους δεν είναι αποτελεσματικά, με αυτές διακόπτουμε τη συνεργασία. Και είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να διασπαθίζουμε το δημόσιο χρήμα. Πολλό δε μάλλον που αντιμετωπίζουμε παντού περιορισμούς και στενότητα οικονομική. Γι' αυτό και το θέμα της λογοδοσίας όλων των εταίρων μας είναι σοβαρότατο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Και την Κυριακή αφιέρωσα δύο ώρες και με ένα επιταλείο που ασχολείται με το θέμα ε, τη, των λογιστικών στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για να ενημερωθώ για αυτά τα θέματα των λογιστικών και απόδοσης λογαριασμών και ευθυνών. Σας ευχαριστώ που θέσατε και τη σχετική ερώτηση. Υπάρχει και συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Μακλάρκιν. Μάλιστα. Έχετε πολύ μεγάλο κύρος από το προηγούμενο σας έργο στην Παγκόσμια Τράπεζα. Φαντάζομαι ήταν απρόσμενος για σας ο διορισμός της υποψήφιας επιτρόπου, ως υποψήφιας επιτρόπου. Γιατί θέλετε να αναλάβετε αυτό το έργο της Επιτρόπου. για δύο λόγους. Καταρχήν ε, είχαμε κάποιες ασυνήθιστες περιστάσεις εδώ και οι συμπολίτες μου, οι συμπατριώτες μου ε, δυστυχώς βρέθηκα σε δύσκολη, δυσάρεστη θέση. Η κόρη μου διαμένει στη Βουλγαρία, η οικογένειά μου το ίδιο και όταν με κάλεσαν το αισθάνθηκα ως καθήκον μου να ανταποκριθώ. Αλλά υπάρχει και το θέμα της τύχης. Υπάρχουν 26 χαρτοφυλάκια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τέσσερα το περιβάλλον, ε, κλιματολογικές δράσεις, ε, ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη είναι τα πιο προσφυλή για μένα. Και ήταν τέσσερα από τα 26 χαρτοφυλάκια που με ενδιέφεραν. Και πραγματικά ήταν ε, σημαντική τύχη. Και ελπίζω, αν με εγκρίνετε κι εσείς, να μπορέσω να αναλάβω αυτό το καθήκον. Σα de κυρία Τσίμερ ευχαριστώ. Κύριε έχετε από την εργασία σα στην ε, Διεθνή Τράπεζα εμπειρίες που θα μπορούσαν να μα χρησιμεύσουν και εδώ. Γιατί η Διεθνή Τράπεζα ήταν ε, η πρώτη οργάνωση που ε, κατέληξε σε πιο ευρία έννοια της και που συνεδίασε την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναεπενικοδόμηση. Από την ιδέα αυτή θα έχετε μια βάση της εργασίας σας όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, βοήθεια ανοικοδόμησης να βασιζόσαστε κυρίως στις ανάγκες των εκεί πολιτών και των περιφερειών και να μην αφήσετε να σας επηρεάσουν τα συμφέροντα την επιχειρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να ωφεληθούν. Ε, η υποψήφια έχει το λόγο. Καταρχήν, ο σύνδεσμος της ανακούφισης, της ε, ανασυγκρότησης ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης δεν είναι αυτόματος πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση. Μερικές φορές δεν φτάνουμε καν στο σκέλος της ανάπτυξης, δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Και σκέφτομαι και το Σουδάν. Μακάρι να μπορούσαμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και στο Σουδάν ή στη Ζιμπάμπουε. Γιατί να αντιμετωπίζει η χώρα αυτή την κατάσταση που βιώνει σήμερα. Αλλά αυτές ευτυχώ είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι ότι πολύ συχνά, πολύ πιο συχνά μπορούμε να εθετήσουμε αυτήν την ολιστική προσέγγιση και να έχουμε όλες τις φάσεις, την ανακούφιση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη. Λυπούμε, αλλά δεν άκουσα και το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Αν κατάλαβα πάντως καλά, με ρωτήσατε πώς αντιλαμβάνομαι το ρόλο των επιχειρήσεων σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι φορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Πέραν των προαιρετικών συνεισφορών και των φιλανθρωπικών δωρεών, δεν βλέπω άλλο ρόλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή συνεργασία, όταν υπάρχει μια πλατφόρμα για ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα και μεταφορά επιχειρήσεων, είναι καλό. Τώρα, όταν έχουμε τέτοια προγράμματα στην τράπεζα, θέλουμε να εξασφαλίζεται σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να πληρούνται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια της Παγκόσμιας Τράπεζας και προωθούμε και στο τραπεζικό κλάδο. Δυστυχώς ε, η πρόεδρος διέκοψε πάλι με το κουδούνι. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, έχω μια συμπληρωματική ερώτηση και αναφέρομαι εδώ στις ε, επιχειρήσεις που δρούν μέσα στα πλαίσια της ε, ανοικοδόμησης ε, και που εκμε... οφειλούνται από το γεγονός ότι υποστηρίζουν τις εργασίες τους με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά με ενδιαφέρουν και οι περιεθνικές ε, επιχειρήσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που με την δική σας βοήθεια είναι υπεύθυνε για κάποιες καταστροφές φυσικών περιφερειών κλπ. Ε, προτίθεστε να ρίξετε τις ευθύνες στις επιχειρήσεις αυτές. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό κλάδο σε θέματα ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική. Αλλά αρμόδιος για τα θέματα αυτά είναι ο Επίτροπος Ανάπτυξης, γιατί εκεί εντάσσονται οι αναπτυξιακές επενδύσεις, στο δικό του χαρτοφυλάκιο. Πάντως, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι έχουμε υποχρέωση να θεσπίσουμε υψηλές προδιαγραφές και η ανάμειξη των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές όντως να προαγάγει καλύτερες ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές καταστάσεις. Ο κύριος Μάριο Μποργέζη. Κύριε υποψήφι Επίτροπε, δείχνετε μεγάλη εμπιστοσύνη στον έλεγχο που ασκεί η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην χρήση αυτών των τεραστίων ποσών που χρησιμοποιεί για την βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω διαφορετική άποψη και θα ήθελα να ξέρω αν δεσμεύεστε να ελέγξετε τους ελεγκτές, να επαληθεύσετε μέσω ελέγχων ε, και στις ε, χώρες δικαιούχους της, βοή... της ενισχύσης αυτές που πάνε και τι γίνονται, γιατί για παράδειγμα κάποιοι οι, οι στην Αφρική μας δίνουν ε, πολύ αρνητικά σημάδια σε σχέση με την ασφάλεια της χρήσης των ποσών αυτών. Και έπειτα η ερώτηση για το ρόλο της στρατιωτικής παρέμβασης. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. So on uh, would I, uh, uh, Δύο ερωτήσεις. Το πρώτο, ψηλά επίπεδο ε, ελέγχου στα οικονομικά. Φυσικά είμαι, με, είμαι υπέρμαχος της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Στην πρώτη μου θέση ε, εργάστηκα για το περιβάλλον γιατί κάποιος ε, πολύ κοντινός μου άνθρωπος ε, αρρώστησε πάρα πολύ βαριά λόγω δηλητηρίασης από βρώμικο νερό το οποίο ήταν υποτίθεται πόσιμο. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει διαφάνεια μπορεί κανεί να πεθάνει. Και για μένα αυτό έγινε δίδαγμα. Ε, θα πρέπει λοιπόν, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, να τους οικοδομήσουμε. Τούτου λεχθέντω, έχω την εντύπωση ότι στο βαθμό που η ανθρωπιστική βοήθεια δίνεται όχι μέσω των κυβερνητικών ε, καναλιών αλλά σε, συνεργα... σε, σε οργανισμούς εταίρους όπως ο, Λευκο... ο Ερυθρός με μεγάλη παράδοση και εντυμότητα, ε, πιστεύω πως αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια διοχετεύεται σωστά και πιστεύω ότι χρησιμοποιούνται οι πόροι μας σοφά. Για το δεύτερο σας ερώτημα, ε, η άποψη της κοινότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, έχει την άποψη πως η στρατιωτική παρέμβαση είναι το τελευταίο καταφύγιο και ότι θέλουν να γίνεται διαβούλευση για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση ή όχι κάθε φορά. Ε, ομολογώ πως πρέπει να μάθω περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα, αλλά από τα όσα έχω μάθει μέχρι στιγμής... Πιστεύω πως είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Διακόπτη πρόοδος. Έχετε μία επερώτηση. Θα δώσω αμέσω στην Επίτροπο την δυνατότητα να συνεχίσει την πρότασή τη, γιατί πιστεύω και θα ήθελα να μα δώσετε την άποψή σα πω αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Δεν είναι, το ουσιαστικό επιχείρημα δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί από τεχνοκρατική άποψη. Το βλέπουμε ότι προέρχεστε από την Παγκόσμια Τράπεζα και εγώ μιλάω για το ευρωπαϊκό δόγμα ενισχύσεων. Θέλετε, θα, θα, καλέσετε εμπειρογνώμονες, θα, θα εμπλέξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε επιτέλους να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δόγμα για τις ενισχύσεις. Σαφές. Η υποψήφια επίτροπος να ολοκληρώσω το θέμα της θεωρητικής παρέμβασης. Έχω ε, την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανθρωπιστική βοήθεια και μέσω αυτής η κοινότητα έχει τη δυνατότητα να το συζητήσει με τους Υπουργούς Αμήνης και τους Υπουργούς Εξωτερικών με κάποιο τρόπο για να δούμε ποια είναι κάθε φορά ο καλύτερος τρόπος. Θα επανέλθω μόλις ε, θα είναι καλό, μόλις θα ξέρω περισσότερα, αλλά σίγουρα η κυρία Άστον θα είναι γέφυρα για την κοινότητα των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών ε, Αμήνης. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ο κύριος Φρανκ Φαν Χέκε, μη γεγραμμένος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, εσείς αναμφίβολα θα γνωρίζετε πως ε, ο Καρλ Ντεγκούχτ ε, ανακηρύχθηκε περσόνα κράτα στο Κονγκό γιατί έκανε δηλώσεις σε σχέση με την πλήρη πτώχευση και αποτυχία του κράτους και της πολιτικής παρά τα εκατομμύρια εκατομμυρίων που έχουμε δώσει στο Κονγκό ακριβώς για να οικοδομήσει το κράτος δικαίου και για να ε, στην ουσία για να στηρίξουμε το, ένα κράτος και να το χρηματοδοτήσουμε. Και τώρα σας ρωτώ, συμμερίζεστε αυτήν την άποψη και πώς ε, θα διαχειριστείτε τις σχέσεις με την κογκολέζικη κυβέρνηση. I think that, that uh, reaching a point when the uh, uh, channels of communication are completely uh, broken is really... Πιστεύω πως ε, όταν ε, διασπώνται οι αυτό είναι πραγματικά λυπηρό, αλλά κάποιες φορές συμβαίνει. Θα έλεγα ότι όσο είναι δυνατόν προσπαθούμε να διατηρούμε έναν δρόμο διαλόγου έναν διεύλο διαλόγου που θα μας διευκολύνει να προχωρήσουμε. Το είδαμε αυτό, το είδαμε και στην Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί ορισμένες φορές ε, κάνουμε το τελευταίο βήμα πολύ αργά. Ε, θα έπρεπε δηλαδή να είχαμε σταματήσει ένα βήμα νωρίτερα. Και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα προσπαθήσω να ενημερωθώ όσο γίνεται καλύτερα. Ε, πιθανότατα θα επανέλθω εδώ, διότι αυτή η Επιτροπή έχει το πλεονέκτημα πέρα από την ε, πολιτική πτέρυγα του καθενός για τις πολιτικές πεπιθέσεις. Έχετε όλοι ένα στόχο, δηλαδή την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Θα επανέλθω εδώ, είναι πολύ δύσκολα σε φάσεις, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν κρίσεις και βασίζομαι και στη δική σας σοφία. Αλλά για να είμαι πολύ κατηγορηματική, εάν έχουμε εξαντλήσει κάθε ε, δυνατότητα συζήτησης και διαλόγου, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, δυστυχώς. Dank u mevrouw, maar vindt u niet dat we eh, toch principiëler moeten zijn en dat wij... Επιρώτηση ο κ. Φανχέκερ. Ναι, ευχαριστώ, αλλά δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια θέση αρχή με βάση την οποία πέρα από τι ανθρωπιστικέ βοήθειε όλε οι ενισχύσει για οι αναπτυξιακέ προ το Κονγκό αλλά και σε άλλε αφρικανικέ χώρε, θα πρέπει να υπόκειται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσπρόοδο όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και την ανοικοδόμηση κράτου δικαίου γιατί χωρίς τέτοια απόφαση επί της αρχής το πρόβλημα δεν θα πάψει. Η υποψήφια επίτροπο. Κοιτάξτε, προσέξτε, γιατί στον τομέα των ευθυνών μου, εάν ε, με εγκρίνετε σε αυτή τη θέση τη ε, ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να είμαστε ουδέτεροι. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι φτάνουμε στον κόσμο. Δηλαδή, η εστίασή μας είναι στο διεθνή ανθρωπιστικό, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και πρέπει σε αυτόν τον στόχο να ε, εστιάζουμε την προσοχή μας. Τώρα, γενικότερα, εκτός αυτού του χαρτοφυλακίου, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, ναι, είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς αρχές. Και πιστεύω τουλάχιστον για μένα, αυτό που με κάνει περήφανη που είμαι Ευρωπαία είναι ότι έχουμε αξίες και τα καταφέραμε δύσκολα. Δεν μας ε, ήρθαν ε, ουρανοκατέβατες οι αξίες αυτές. Στην Επιτροπή περιβάλλοντος ε, ε, έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, οι φυσικές καταστροφές, οι φυσικές θεομηνίες κλιμακώνονται τα τελευταία χρόνια και οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές, το γνωρίζουμε αυτό. Στην Ευρώπη έχουμε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Στην Νότια Ευρώπη έχουμε εκατοντάδες ε, εκτάρια που καταστρέφονται τις κάθε χρόνο. σε πολλές περιπτώσεις οι δυνατότητε των κρατών μελών να ανταποκριθούν είναι ακατάλληλε λόγω του μεγέθους των φαινομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το περασμένο καλοκαίρι ζήτησε την ενίσχυση της, ε, των δυνατοτήτων ε, προστασίας των πολιτών ε, της κοινότητας. Θα απαντήσετε θετικά σε αυτό το αίτημα. Πώς θα το κάνετε αυτό, εάν προτίθεστε να το κάνετε. Υποψήφια Επίτροπος, δύο λεπτά. Με την προστασία των πολιτών που προέρχεται από το Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στην ε, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα έχουμε μια νέα οπτική και θα προετοιμαστούμε για τον επόμενο κύκλο, ίσως να μην χρησιμοποιώ το σωστό όρο, με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει για την επόμενη μας φάση, όταν θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, και είναι πολύ κέρια στιγμή. Ε, θα σας πω ότι είμαι πεπισμένη γιατί προσωπικά πιστεύω στην ανάγκη να είμαστε έτοιμοι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ε, ήμουν διευθύντρια της Παγκόσμιας Τράπεζας στη Ρωσία, Συνεργαστήκαμε με τη ρωσική κυβέρνηση για να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό των μετρολογικών υπηρεσιών τους. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση για τη Ρωσία τώρα, αντιμετώπιζε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και οι Ρώσοι για να αναγκαστούν να δανειστούν από την Παγκόσμια Τράπεζα για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις μετρολογικές υπηρεσίες δεν ήταν πολύ προφανές. Κάναμε λοιπόν μια οικονομική ανάλυση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και τώρα θα σας αναφέρω ένα μέτρο από το οποίο χρησιμοποίησαμε τότε. Τι κάναμε. Ε, συμπεράναμε ότι για κάθε δολάριο που δαπανίσαμε για τις μετεωρολογικές υπηρεσίες είχαμε κέρδος 16 δολάρια από τις προληπτικές δράσεις. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πεποίθησή μου, γιατί οι αποδείξεις είναι συντριπτικές ότι η πρόληψη είναι η πιο σημαντική και η ετοιμότητα είναι πολύ κρίσιμη και από μόνη της ωφελεί και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Μόλις θα γίνει λοιπόν η αναθεώρηση και θα δούμε τι δεν είναι σωστά ε, προγραμματισμένο, φυσικά και θα προβούμε σε δράση. Θα επανέλθω εδώ στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα. Και τώρα έχουμε το δεύτερο γύρο. Α, συγγνώμη, έχετε επερώτηση. Είπατε αναθεώρηση. Υπήρξε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το περασμένο καλοκαίρι. Ε, υπήρξαν κάποια ευρωπαϊκά ε, πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πολύ χρήσιμα ήταν θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ή θα σταματήσει φέτο το καλοκαίρι. Εγώ δουλεύω για αυτό το πρόγραμμα, το είδα, το διάβασα συγγνώμη και είδα ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό τώρα που δεν είναι σαφές είναι αν θα συνεχίσουμε, αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική κατάσταση, δεν ξέρω πού μπορούμε να βρούμε χρήματα για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα γιατί κλείνει το 2010, αλλά ελπίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να το συνεχίσουμε, γιατί... Τουλάχιστον μία φορά τελείωσα στην ώρα μου, κυρία Πρόεδρε. Ναι, πάντως, αν μπορέσουμε να βρούμε χρήματα, θα το συνεχίσουμε. Δεύτερος γύρος ερωταπαντήσεων. Το λόγο έχει ο κύριος Κατσμάρεκ. Ε, Ευχαριστώ. Στην εισαγωγική σας ομιλία, κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Συνένεση σε θέματα ευρωπαϊκής ενίσχυσης. Το 2008 θεσπίστηκε το πρόγραμμα δράσης για τη συνένεση αυτή. Ερωτώ. Θεωρείτε ότι αυτά τα σχέδια δράσης είναι σημαντικά και έχουν προτεραιότητα και για σας. Όταν το επιτελείο της ε, Γενικής Διεύθυνσης με ενημέρωσε, εντυπωσιάστηκα γιατί υπάρχουν 49 προγράμματα και στα 42 έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Από τους τομείς δράσης, δύο ξεχωρίζουν κατά την άποψή μου, που θα, ελπίζω πως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Το ένα είναι ο συντονισμός και φυσικά δεν θα σας εκπλήξει, δεδομένης της συζήτηση που σήμερα, που έχουμε σήμερα. Και το δεύτερο είναι η συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων και φορέων. Ευχαρίστω θα επανέλθω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Αν με εγκρίνετε βέβαια. Μόλις θα έχω πιο σταθμισμένη άποψη. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες στην ερώτησή σας. Συμπληρωματική ερώτηση θα γίνει κάποια αναθεώρηση αυτών των σχέδιων δράσης φέτος. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. This, this is correct. That's very true. Yeah. Ναι, ναι, σωστά. Δώστε μου λίγο χρόνο να προετοιμαστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πατρίς Τερολία. Ε, madame, euh, dans vos réponses, Κύριε Πρόεδρε, μετά από την καταστροφή αυτή στην αιτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε δυνατότητα να αντιδράσει όσον αφορά το σε κατάσταση του ανθρωπίνου Οι προσπάθειε του νοσμού τη κυρία Άστον είναι αξιόλογε, αλλά οι μεμονωμένε αντιδράσει δεν είναι ε, ισότιμε με τι οργανωμένε απαντήσει των Ευρωπαίων. Είδαμε πολλέ απαντήσει που οδήγησαν σε μια έλλειψη ορατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επιτόπου. Εσείς θα φροντίσετε να υπάρχει συντονισμένη ε, αντιμετώπιση και ότι να είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο ακριβή. Η υποψήφια αντιεπίτροπος έχει το λόγο. Το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας χρησιμοποιείται κατά βάση πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αλλά έχουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Τα τελευταία δέκα χρόνια, από τα τελευταία 10 χρόνια, κατά διάρκεια των 9 ετών, τα χρήματα που δόθηκαν μέσω αυτού του μέσου δεν ήταν επαρκή. Και όταν χρειαζόταν περισσότερο χρήματα, ε, λήφθηκαν από την Κομισιόν. Αυτό κατά με είναι μια ένδειξη αυτού που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ότι αυξάνεται ο αριθμός και η ε, σοβαρότητα των ε, ε, φαινομένων που οδηγούν στην ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι και άλλα μέσα της Κομισιόν έχουν χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθούν εκείνοι που βρίσκονται σε κάποια κατάσταση ανάγκης, παραδείγματος μέσα στα πλαίσια της τη Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης δίνει 150 εκατομμύρια ευρώ, αν χρειαστούν, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και τελευταία έχουν ήδη ληφθεί από εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι όποτε χρειάζεται έχουν κινητοποιηθεί οι διάφοροι πόροι. Και τα κρατημέλα βέβαια βοηθούν στις περίπτωση ανάγκης. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ε, πιο ικανοί, πιο καινοτομικοί όταν χρειαστεί να κοινοποιήσουμε κάποιους πόρους. Παραδείγματο χάρη και είμαι περήφανη αυτό από την εργασία μου στην ε, Διεθνή Τράπεζα. Είχαμε μια ιδέα για την ασφάλιση ε, καταστροφών για πολύ φτωχέ χώρε. Και η παραδείγματο χάρη η Χαϊτή είχε μια τέτοια ασφάλεια που πλήρωσε η καναδική κυβέρνηση τα ασφάλιστρα για 300, 300 εκατομμύρια και την επομένη της καταστροφής αυτά τα χρήματα διατέθηκαν καταρχήν. Μπορούμε έτσι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο εύκολα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Πρόταση πρέπει να συνεχίσουμε. Και ίσως δεν υπάρχει και συμπληρωματική ερώτηση. Το λόγο κύριο Σίβε Μπάγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργίευα, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για τον ε, ήπιο τρόπο και με τον οποίο εδώ και για τις ικανότητες που διαφαίνονται να έχουν. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για, τους ανθρωπογενείς, ε, για τις ανθρωπογενείς καταστροφές, ε, δηλαδή καταστροφές οι οποίες δημιουργούνται από στρατιωτικές παρεμβάσεις των γειτονικών χωρών. Στην δηλαδή, με τους χάρη. στις καταστροφές αυτές πλήττεται κυρίως ο άμαχος πληθυσμός. Και στην περίπτωση θα πρέπει οι χώρες να λάβουν υπόψη τους περισσότερο την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και σταθερότητας. Συμφωνείτε μαζί μου, θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Η υποψηφία επίτροπος έχει το λόγο. Θα ήθελα να επανέλθω στις αρχές σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται η ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίοι απαινούν ουδετερότητα και ανεξαρτησία για τους ε, εργαζόμενους στα πλαίσια της βοήθειας. Η κυβερνήση λοιπόν συχνά δεν είναι η σωστή διαβλός δράσης. Ξέρουμε βέβαια πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν ε, χώρε οι οποίες είναι πάρα πολύ ευάλωτε ή που έχουν αποτύχει ω κυβερνήσει. Εγώ δεν νομίζω θα είναι δική μου ευθύνη να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, αλλά όπως είπα και εισαγωγικά, <clears throat> να πρόκειται να αναμετωπίσουμε αδικίες εις βάρος των πολιτών ή πληγές κατά των παιδιών των γυναικών θα υψώσω τη φωνή μου. Θα κάνω λόγω της θέσης μου ό,τι μπορώ για να υψήσω την προσοχή στο συγκεκριμένο πρόβλημα, στις απαράδεκτες αυτές τις καταστάσεις και συμπεριφορές. Ίσως δεν κατανόησα όλοι σας την ερώτηση, γιατί κάποιο, κάποια φασαρία άκουσα εδώ, κάποιο θόρυβο και ίσως δεν σας άκουσα καλά. Ίσως αν δεν σας απάντησα σωστά, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, συμπληρωματική. Όχι, είναι ένα σχόλιο, δεν είναι ερώτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την, ερώτηση, για την απάντηση που δώσατε, που ήταν πάρα πολύ καλή και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε ένας να χρησιμοποιήσετε πραγματικά όλη σας ε, την ε, ισχύ για να φτάσετε πραγματικά να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που έχετε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας η υποψήφια επίτροπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Ο κύριος Πατστάς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε. Γνωρίζετε την κατάσταση στην Γάζα. Η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί είναι φοβερή. Ε, το Ηνωμένο Έθνη και η ΟΥΝΤ να λένε ότι 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση εκεί. Πώς θα φροντίσετε με τους 26 ε, επιτρόπους ε, συναδέλφους σας να πίεσετε το Ισραήλ να επιτρέψει κοβά ανθρωπιστικά να περνάμε και τι θα κάνετε για να μην συνεχίσει να βρίσκεται στην κατάσταση αυτή η Γάζα απάντηση. Πραγματικά εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο θέσατε την ερώτησή σας. Είπατε τι θα κάνω μαζί με τους 26 συναδέλφους. Ναι, προφανώς. Η προσέγγιση θα πρέπει να είναι μια συλλογική προσέγγιση. Εγώ από πλευρά μου έχω να πω ότι αυτό πραγματικά που προβληματίζει τους επιτόπου εργαζόμενους είναι το θέμα της πρόσβασης. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ περιορισμένη είναι τώρα στο 20-25% από ό,τι ήταν πριν από το 2006. Το πιο σημαντικό για μας είναι να ζητάμε και να επιμένουμε πρόσβαση. Αλλά πώς θα γίνει αυτό. Επιζώντας την προσοχή, ναι. Αλλά και συνεχώς χτυπώντας τους λόγους για τους οποίους λέγεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης. Από ό,τι κατάλαβα παραδείγματος χωρίς ένας λόγος που αναφέρεται είναι ότι ίσως ορισμένα τα αγαθά που μεταφύγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς λόγους. Ωραία. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή και το κάνουμε νομίζω. Να τους πούμε. Δώστε μας ένα αρνητικό κατάλογο να μας πείτε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό δεν επιτρέπεται να περάσει ή δώστε μας ένα θετικό κατάλογο που να λέει αυτά μπορείτε να τα περάσετε στην Γάζα. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα, το πρώτο είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ενωμένη, να μιλήσουμε με μία φωνή και δεύτερον να καλύψουμε όσο μπορούμε τους επιτόπου εργαζόμενους και να άρουμε θεωρητικά ή πραγματικά τεχνικά εμπόδια. Συμπληρωματική ερώτηση κύριε Αμπάρτς. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την ε, απάντησή σας και θα ήθελα να πω και το εξή ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συμφωνίες συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ όπου προβλέπεται ανοιχτή πρόσβαση του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτέ τι συζητήσει, ούτω ώστε το Ισραήλ να αναγκαστεί να αναλάβει θετικέ δράσει προ την κατεύθυνση αυτή. Υποψήφια Επιτροπή, ναι, μα ακριβώ γι' αυτό τόνισε αυτό το σημείο τη της ε, ερώτηση Θα πρέπει να δούμε το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουμε με το Ισραήλ. Εγώ δεν μπορώ να σας πω κατά πόσον αυτό γίνεται, πώς πρέπει να γίνει, αλλά οπωσδήποτε αυτό το μήνυμα θα το περάσω στο συλλογικό όργανο των επιτρόπων και αυτό είναι το έργο μου να ε, φροντίσω να καταλαβούν όλοι ότι υπάρχει μια κρίση και πρέπει κάτι να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ντέβα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπα ψήφια, Επίτροπε. Θα είσαστε, είπατε, η φωνή εκείνο που δεν έχουν φωνή. Τελευταία προσφυγή εκείνο που μένουν πίσω θα πρέπει να προωθηθεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωση Ο κ. Πίπερ θα αναφέρεται στο εμπόριο. Εσεί, θα μιλήσετε υπέρ εκείνων που είναι άφωνοι, που δεν έχουν φωνή. Θα πρέπει να ε, καμιά φορά να έρθετε σε αντιμέτωπη με, ε, συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωση σε Ναι, ναι, μάλιστα. Έχετε συμπραγματική ερώτηση, λέει η πρόεδρος. Όχι, μετά από αυτή την απάντηση όχι. Ελπίζω όμως και οι άλλοι επίτροποι να σας ακούσουν. Μετά από το σεισμό στην ε, Αϊτή, η ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και γλίγορα και υπήρχε συντονιστό των εθνικών ε, μέσων. Είπατε ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι, ποια είναι που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Ποια είναι τα μέτρα που προβλέπετε εσεί για να βελτιωθεί ο συντονισμό, η συνοχή και ε, ανασύνδεση, Ποιο θα είναι, θα είναι ο ρόλο τη ομάδα εργασία ΚΟΑΦΑ και ε, επιστημονική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία μια ευρωπαϊκή δύναμη προστασία των πολιτών θα είναι μία από τις προτεραιότητές σας και πώς θα οργανωθεί αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η υποψήφια επίτροπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. <clears throat> Πράγματι, το γεγονός ότι υπάρχει επίτροπος για τον διεθνή συντονισμό και την ανθρωπιστική βοήθεια είναι ήδη ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση και ξέρω ότι υπάρχουν δύο ομάδες στο Συμβούλιο, η ΚΟΧΑΠΑ όπως είπατε, που ασχολείται η μία με την ανθρωπιστική βοήθεια και με την επιστική βοήθεια και η ομάδα πρόσεκ που ασχολείται με την προστασία των πολιτών και θα είναι σίγουρα απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο μέθοδοι και να δούμε εάν υπάρχει κάποιο ανάγκη συγχρονισμού των δύο για να κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα του, της Χαϊτής για να προχωρήσουμε προς το προς. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά το τσουνάμι υπήρχε μια πολύ καλή αξιολόγηση που έγινε για τα διδάγματα από το τσουνάμι. Κοιτάμε τώρα στην ΑΕΤ και βλέπουμε ότι ορισμένα από αυτά τα διδάγματα πραγματικά εφαρμόστηκαν. Σε μεγάλο ποσοστό. Όχι όλα, και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δάγματα στα οποία καταλήγουμε από την IT. Θα πρέπει να δούμε τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε τόσο σωστά και πώς θα μπορούμε να βελτιώσουμε. Και νομίζω ότι στις ε, δύο αυτές ομάδες του Συμβουλίου έχουμε ήδη την πλατφόρμα για να αποχωρήσουμε με τα κράτη-μέλη και βέβαια στην συνεργασία με τη δική σας εδώ Επιτροπή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Γιώαν Πάσκου. Ένα λεπτό κύριε Πάσκου. Well, I have a problem because I had two... Έχω ένα πρόβλημα γιατί είχα προετοιμάσει δύο ερωτήσεις αλλά με πρόλαβαν οι συνάδελφοι και όχι μόνο τις ε, υπέβαλαν αλλά τις απαντήσατε κιόλας. Έχουμε ένα θέμα που είναι πολιτικά πολύ φορτισμένο. Πώς θα συνδυάσετε την ανάγκη άμεσης δράσης αφενός με την μακροπρόθεσμη προοπτική που έχει κατά ανάγκη η πολιτική δράση. Πώς θα τα συμφιλιώσετε αυτά τα δύο. Για την ανθρωπιστική βοήθεια, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ταχύτητα η αμεσότητα. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί γρήγορα, να φτάσει ταχύτατα στους αναξιοπαθείς, αυτούς που τη χρειάζονται. Αυτή η ανάγκη για μας είναι ο κινητήριος μοχλός. Η ανάγκη της ταχύτητας. Τώρα, αν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, όπως δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά, όπου η ανασυγκρότηση, η ανοικοδόμηση και η ανάπτυξη δεν είναι φάσεις που ακολουθούν της ανακούφισης, τότε έχουμε πρόβλημα. Και δημιουργείται μια μακροχρόνια παράδοση εξάρτησης από τη βοήθεια. Και έτσι χάνονται ζωές, ε, διακυβεύεται το μέλλον των ανθρώπων, ε, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το παραγωγικό τους δυναμικό, δεν μπορούν να ξαναβρούν δουλειά. Όσο διαιωνίζεται αυτή η φάση της εξάρτησης από την ανθρωπιστική βοήθεια, τόσο πιο δύσκολη είναι η επαναφορά στην ανοικοδόμηση και στην αναπτυξιακή φάση. Εκεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε την πολιτική μας κρίση και να δούμε πότε έχουν οριμάσει οι πολιτικές προϋποθέσεις. Γιατί αν παρά είναι υψηλές οι προδιαγραφές και οι απαιτήσει μας, τότε ίσως έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορούμε να, ε, αντί να βοηθήσουμε, να βλάψουμε περισσότερο τον κόσμο. Βέβαια, τέτοιου είδου κρίσει προποθέτουν όχι μόνο μια ορθολογική πολιτική αξιολόγηση, αλλά και μια συναισθηματική αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν ανοιχτές και διαφανείς πληροφορίες, ώστε να έχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε γνώμη με όσο το δυνατό πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο. Υπάρχει επερώτηση για το θέμα αυτό. Όχι, όχι, καλύφθηκα. Ωραία. Προβλέφθηκε και ένα διάστημα για ερωτήσεις που έχουν υποβάλει γραπτός οι πολιτικές ομάδες σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επίτροπο. Έχω λάβει γραπτός λοιπόν διάφορες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Ποια είναι τα διδάγματα που αντιλήσατε από την αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο σεισμό της ΑΕΤΗΣ. Πώς πιστεύετε ότι τα διδάγματα αυτά θα επηρεάσουν ε, τα καθήκοντά σας ε, ως αρμόδιας επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχετε ένα λεπτό να απαντήσετε στην ερώτηση. Και 45 δευτερόλεπτα. Φυσικά θα περάσει η κρίση και θα γίνει μια πιο συστηματική αξιολόγηση των διδαγμάτων που αντλήσαμε από αυτή. Μέχρι στιγμής πάντως έχω τρία σχόλια. Καταρχήν, όσοι έχουν αναλάβει αυτό το έργο βρέθηκαν επιτόπου στην ΑΕΤ, χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν τα διδάγματα από το τσουνάμι. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν κάποια αποθέματα επιτόπου, ώστε να μην ε, πρέπει να τα μεταφέρουμε από την Ευρώπη. Υπάρχουν σε, διάφορα, σε διάφορες τοποθεσίες πιο κοντά και αυτό ήταν, συνέβη και στην ΑΕΤ και ήταν πολύ χρήσιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία για το ποιο ήταν το έργο της Ευρώπης, δεν ήταν αρκετή, γιατί συναντήθηκα με την ομάδα επιτόπου και κάθε μέρα γινόταν αξιολόγηση για το τι συνέβη, ποιε ήταν, ποιες ήταν οι δράσεις και ήταν πολύ εντυπωσιακές οι δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, αλλά δυστυχώς η επικοινωνία δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική και η εντύπωση που δόθηκε δεν ήταν αρκετά σημαντική. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξουμε τη δράση αλλά και την επικοινωνία γιατί αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι αυτό που πιστεύει, όχι αυτό που συνέβη πραγματικά. Δεν ήταν αρκετά ορατή λοιπόν, δεν προβλήθηκε αρκετά η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει καλύτερη ε, ευκαιρία για συντονισμός ώστε να φανεί η ευρωπαϊκή ανταπόκριση και να βελτιωθεί και η επικοινωνία μας, να προβάλλουμε καλύτερα το ρόλο της Ευρώπης και τη συμβολή της Ευρώπης ως ενιαίου φορέα και όχι ως ε, μία επιπλέον οντότητας ε, πέραν των 27. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έστειλαν ένα πλοίο νοσοκομείο στην ΑΕΤ. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Και πάλι είναι θέμα συνεργασίας των ε, στρατιωτικών ε, και πολιτικών επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι η στρατιωτική επιχείρηση είναι η έσχατη λύση που μπορεί να είναι χρήσιμη ίστατο μέτρο μόνο. Όταν είχαμε τις συζητήσεις ε, με το προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και αναλύσαμε αυτό το θέμα, των ρευστών συνόρων μεταξύ της στρατιωτικής απάντησης και της απάντησης πολιτικής προστασίας, ρώτησα, πιστεύετε ήταν σκόπιμο που ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών επενεύει στην ΑΕΤ και είπαν φυσικά. Άλλος τρόπος δεν υπήρχε εκεί. Γιατί δεν υπήρχε το κυβέρνηση ούτε τίποτα στην ΑΕΤ. Οπότε ήταν σκόπιμη η επέμβαση του στρατού. Όταν έχουμε παρόμοιες περιστώσεις ε, με κατάρρευση της κυβέρνησης, η ανύπαρκτη κυβέρνηση και υπάρχει μια θεομηνία καταστροφή, τότε μπορεί να αναλάβει κάποιο ρόλο και ο στρατός. Αλλά με πολύ προσοχή, γιατί από τη στιγμή που αρχίζει μια στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να ανακληθεί. Είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Σχόλιο εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Και τελευταία ερώτηση. Πώς θα εξασφαλίσετε μια πιο προβλέψιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το Σουδάν συγκεκριμένα. Η ανθρωπιστική βοήθεια δίνεται εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Βασίζεται στις ανάγκες. Οπότε ο καλύτερος προγραμματισμός εξαρτάται από τρία πράγματα. Γίνεται μια σωστή αξιολόγηση των αναγκών. Γνωρίζουμε που εντοπίζονται οι ανάγκες. Δεύτερον, έχουμε κινητοποίηση ε, τα μέσα που χρειάζονται για να καλύψουμε τις ανάγκες. Και τρίτον, υπάρχει πρόσβαση. Μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα τρία σκέλη, οι τρεις απαιτήσει. Σε περιπτώσεις έχουμε πρόβλημα πρόσβασης. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε καν να εντοπίσουμε τον κόσμο που χρειάζεται τη βοήθεια. Και σε άλλες περιπτώσεις ε, το προσωπικό μας δεν μπορεί να φτάσει στους αναξιοπαθείς. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε και τα τρία στοιχεία επιμελώς. Να γίνει μια σωστή αξιολόγηση και ακριβής αξιολόγηση των αναγκών, να εξασφαλιστεί η κινητοποίηση των απαραίτητων μέσων γιατί δεν θα πρέπει απλώς να στέλνουμε ότι μας περισσεύει τι έχουμε, αλλά ότι χρειάζεται πραγματικά και φυσικά να εξασφαλίσουμε και την πρόσβαση ώστε να φτάνουμε στον κόσμο που τη χρειάζεται. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που θα πρέπει να επισημανθούν και να τα επεξεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. Περνούμε στο τρίτο γύρο των ερωταπαντήσεων. Το λόγο έχει η κυρία Κορίνα Κρέτσου. Ευχαριστώ. Θα παραμείνω στο ίδιο θέμα. Το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια του προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκεί που υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις, παράδειγμα το Κογκό, ή άλλες περιπτώσεις ε, είχαμε επιθέσεις σε αποστολές ανθρωπιστικές. Και είχαμε και την περίπτωση της ΑΙΤΙΣ πώς ε, θα μεριμνήσουμε για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό και πώς θα ενισχύσουμε την ασφάλεια του προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η υποψήφια επίτροπος. Αυτό που μάθαμε από ανθρώπους που εργάζονται υπό αντίξωες συνθήκες είναι ότι πολύ συχνά προτιμούν να μην τη χάνουν στρατιωτική συνοδείας. Προτιμούν να είναι μόνοι τους και να φτάσουν στον κόσμο. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει και στρατιωτική παρουσία, είναι αμφίβολη και αφισβητήσιμη ουδετερότητα και ανεξαρτησία αυτή τη στρατιωτική παρουσία. Μερικέ φορέ, βέβαια, είναι επιτακτική ανάγκη η παρουσία του στρατού και πριν από λίγο το ανέφερα δική μου δουλειά, δικό μου καθήκον είναι να είμαστε ανοιχτοί και να γίνεται σωστή αξιολόγηση και αντικειμενική αξιολόγηση των περιστάσεων. Κάτι που έμαθα και το έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι στόχος μας στο Κονγκό για παράδειγμα, κυρίως για το Κονγκό εξαιτία των διαστάσεων της χώρας, πολύ συχνά χρειαζόμαστε πτήσεις από το Σουδάν. Και τώρα τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει καλύτερη προστασία για το προσωπικό, να χρησιμοποιηθούν πτήσεις από το Σουδάν αντί να γίνει χερσαία μεταφορά από... σε μια χώρα που υπάρχουν δύσκολες συνθήκες. Προτιμούμε να πετάνε εκεί παρά να πηγαίνουν οδικώς. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η διασύνδεση και επενδύουμε σε τέτοιες υπηρεσίες διασύνδεσης. Και στην IT η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε μια κεραία για να, μπορεί, να μπορούν οι άνθρωποι να τηλεφωνούν στις οικογένειάς τους και να τους λένε ότι είμαι σώος και αυλαβής. Και η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια, αξιολόγηση της κατάστασης ασφάλειας για το προσωπικό τη ανθρωπιστική βοήθεια. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, όλα αυτά που μα λέτε, αλλά κουδουνίζει πάλι η πρόεδρο, Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την επερώτηση τη κυρία Κρέτσου. Okay. Uh, two... Πέρυσι είχαμε πάνω από 200 ανθρώπους προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας που έχασαν τη ζωή, τους, τη ζωή τους. Θα πρέπει να γίνει σωστή έρευνα, διαλεύκανση αυτών των θανάτων και να δοθεί κάποια συνέχεια. Μάλιστα. Το λόγο έχει ο κύριος Μπιλ Νιούτον Ντάν. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κατά τη γνώμη μου τα πάτε πάρα πολύ καλά. Εδώ εξετάζουμε πώς θα, ε, θα επιτελέσετε το έργο σας. μιλάτε άπτωστα, άπτεστα τη Ρωσική. Περάσατε τρία χρόνια στη Μόσχα. Δεν ξέρω αν είναι εκτός ε, της εντολής σας, αλλά ε, πώς ε, θα συνεργαστείτε, πιστεύετε υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τη Ρωσία για το δικό του σκέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχω δύο εμπειρίε από την παραμονή μου στη Ρωσία που θα μπορούσα να τι αξιοποιήσω. Όταν ήμουν εκεί διευθύντρια τη Παγκόσμια Τράπεζα, είχαμε μια ανθρωπιστική επιχείρηση ταυτόχρονα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της, ε, των Ηνωμένων Εθνών για τον Κάφκασο, για την Τζετζενία και τι γειτονικέ δημοκρατίε. Εκεί, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη, παρακολουθήσαμε την κατάσταση ως εξής. Βέβαια, η Παγκόσμια Τράπεζα δεν παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά διευκολύνει την παροχή βοήθειας και χρησιμοποιεί την πρόσβαση που έχουμε στην ηγεσία της Μόσχας και στις αρμόδιες αρχές και των ενδιαφερόμενων δημοκρατιών. Και έτσι, στον Τατζικιστάν, στο Καμπαρδίνο και στις γειτονικές περιοχές ε, διευκολύναμε ακριβώς την πρόσβαση της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Και προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε λογοδοσία της διοίκησης που λάμβανε την ανθρωπιστική βοήθεια για να είναι απρόσκοπτη η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Βέβαια στην Τσετσενία δεν μπορέσαμε να δράσουμε, αλλά φέραμε κάποιους Τσετσένους στο Καμπαρντίνο Βολγάρια για να τους εκπαιδεύσουμε. Και μάλιστα είχα την τύχη ε, να είμαι στη Ρωσία όταν ε, φιλοξένησε το G8. Και μάλιστα με ρώτησαν τι να κάνουμε γιατί ήμουν αρμόδια στα ε, αναπτυξιακά. Είπα γιατί δεν διοργανώνεται και μια συνδιάσκεψη δωρητών, γιατί είστε νέο δωρητή. Προσκαλέστε και τους υπόλοιπους δωρητές. Αν δεν κάνω λάθος αυτό συνέβη τον Απρίλιο του 2004. Δεν θυμάμαι πότε οργάνωσε η Μόσχα το G8. Δυστυχώ πάλι με το κουδούνι η πρόεδρο ε, ε, διακόπτη συμπληρωματική ερώτηση. Καλώ θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Συμπληρωματική ερώτηση που σχετίζεται με την πρώτη ερώτηση του κυρίου Γκάι Μίτσελ. Πώς θα ε, προβληθεί καλύτερα το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως θα μπορούσατε να ανοίξετε ένα blog ή τουλάχιστον οι υπάλληλοι σας και το Twitter, γιατί όχι να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δίκτυα. Νομίζω ότι το Twitter είναι καταπληκτικό για τέτοια περίπτωση. Γιατί με το Twitter δίνουμε και τίτλους ε, για τους δημοσιογράφους για να γράφουν στις εφημερίδες, τα άρθρα τους. Βέβαια, εγώ είμαι της παλιάς γενιάς και δύσκολα παρακολουθώ αυτές τις εξέλιξεις. Πάντως, το Twitter το παρακολουθώ. Και μάλιστα όταν ε, διορίστηκα υποψήφιο χρειάστηκε να ε, συνομιλήσω με την οικογένειά μου γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες από το Twitter και ήθελα να το μάθουν πρώτα από μένα. Είναι πολύ ισχυρό εργαλείο αυτό γιατί είναι σύντομο και όταν κάποιο είναι περιορισμένο ε, είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο αυτό που θα πει και το μήνυμά του είναι πιο πυκνό και μεστό. Το λόγο κυρία Λέβιν για του πρασίνου. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ βρίσκομαι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιες συνέπειες ε, βλέπετε να υπάρχουν ε, μετά από την αποτυχία της ε, Κοπενχάγης όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια λόγω του αυξημένου κινδύνου για θεομηνίες. Η Κοπεχάγη δεν αποτελεί αξιόπιστο τρόπο για το περιορισμό του παγκόσμιας, της θέρμανσης μάλλον του πλανήτη στους δύο βαθμούς. Πώς πιστεύετε πως αυτό θα επηρεάσει την ανθρωπιστική βοήθεια τα επόμενα πέντε χρόνια, πώς θα υπολογίσετε την αύξηση του κινδύνου και όταν, όσον αφορά την ε, πολυεθνική συνεργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες, τι συγκεκριμένα βήματα θα ασκήσετε ώστε οι πολυεθνικές εταιρείες να, να τηρήσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ που χρειάζονται για να προληφθούν οι καταστροφές, η υποψήφια επίτροπος. Ίσως επειδή προέρχομαι από την ε, τον κλάδο του περιβάλλοντος, να σας πω ότι ήμουν στην Κοπενχάγη και εγώ είχα ανάμεκτα αισθήματα. Δεν ήμουν μόνο αρνητική. Ήταν προβληματικό το θέμα, ήταν πολύ χαοτική η κατάσταση και ήταν και πρόβλημα ότι από την Ευρωπαϊκή Άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν ε, κατάφερε να έχει την θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό θα πρέπει επίσης να το σκεφτούμε στη συνέχεια αλλά πριν από πέντε χρόνια Δεν, θα, δεν περίμενα ότι θα δούμε 120 επικεφαλής ε, κρατών και κυβερνήσεων να βρεθούν στον ίδιο χώρο για να συζητήσουν τις κλιματικές αλλαγές. Ήδη αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση. Νομίζω πως έχει ε, βελτιωθεί η κατάσταση στην Κο, Κοπενχάγη για τους 40.000 ανθρώπους εκεί και το χάος και αυτό βοήθησε στην συνειδητοποίηση και στη γνώση. Δηλαδή δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία. Για την ερώτησή σας, ε, συμφωνώ πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση των ε, καταστροφών. Κάτι για το οποίο δούλεψα στην τράπεζα ήταν ο βάλτος χαρακτήρα των φτωχών χωρών απέναντι στις κλιματικές αλλαγές. Και το θέμα είναι, θα σωρεύσουμε πόρους ή θα βρούμε δραστήριους τρόπους για να κινητοποιήσουμε τους πόρους αυτούς. Θα πρέπει δηλαδή να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο γιατί αν πιστεύουμε πως με τους προϋπολογισμούς βοήθειας θα γλιτώσουμε τον κόσμο και τις χώρες μετά από 10-15 χρόνια δεν θα μπορούμε πια να το κάνουμε. Άρα λοιπόν η δουλειά μου είναι να συνεργαστώ, η πρόεδρος διακόπτη με το καμπανάκι της. Έχετε περώτηση Μπορείτε να επεκταθείτε κάπως στο πώς θα μπορέσετε να επηρεάσετε τους πολυεθνικούς ομίλους στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές για το περιβάλλον. Ξέρετε, Κοιτάξτε, δεν είναι και εκεί όλα μαύρα. Υπάρχουν εταιρείε που ε, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και έχουν αναλάβει την ευθύνη για όσου εργάζονται στην, χώρα, στην ε, εταιρεία μέσα στι αναπτυσσόμενε χώρε και δεν είναι τόσο μειοπικέ Όλε. Υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορούμε όλους να τους βάλουμε στο ίδιο καλάθι και να τους διαγράψουμε εγώ μπορώ να πω ότι πολύ υπεύθυνα πως πολλές εταιρείες έχουν αντιδράσει θετικά. Μα κάποιες όμιλοι είναι πολύ ισχυρότεροι και μεγαλύτεροι από τις ίδιες τις χώρες. Έχουν ευθύνες και οι ίδιες. Πώς μπορούν οι πολίτες να στηρίξουν το... Διακόπτη πρόεδρος. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Εύα Σανίκινη. Πίσω σας, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπο. Θα πρέπει να σας πω ότι πολύ μου αρέσετε, γιατί είστε ε, γυναίκα με κλάση και είστε πολύ σαφείς και ξεκάθαροι στα όσα μας λέτε και πολύ ειλικρινείς. Ε, με τον κύριο Επίτροπο Ντεγκούχτ μετά την ΑΕΤ, η Amnesty International και άλλε ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις κατήγγυλαν την εξαφάνιση δεκάδων παιδιών που γλίτωσαν από το σεισμό. Και ε, επέσαν την προσοχή του Επιτρόπου στου τεράστιου κινδύνου κατάχρησης και παράνομων εμπορίων των ανηλίκων. Ποιες, με, ποια μέτρα έχουν ληφθεί λοιπόν ή σκοπεύετε να λάβετε για να παρακολουθήσετε και να προστατέψετε αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Very encouraged that UNICEF is taking on this issue very seriously. UNICEF ασχολείται με το θέμα πολύ σοβαρά. Έχουν δώσει πολλές πληροφορίες που μας βοηθούν πάρα πολύ ώστε να μπορέσουν όλοι να σχηματίσουν γνώμη για το θέμα. Και όταν λέω οι άλλοι, εννοώ ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις. Γιατί κατάλαβα ότι τμήμα των ε, υιοθετήσεων που είχαν ήδη νομικά, νόμιμα μάλλον συμφωνηθεί πριν να χτυπήσει ο σεισμός, ένα τμήμα είναι οι καλοί άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά ένα άλλο τμήμα είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να οδηγήσει όντω στην εμπορία παιδιών. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πω, όπω και άλλοι στην UNICEF, και να, να μιλήσω γι' αυτό, να γίνει γνωστό, το κοινοβούλιο να γνωρίζει τι συμβαίνει, ότι δηλαδή ε, πάει αυτό στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Όσοι δηλαδή μπορούν να βοηθήσουν να, μπορούν να, το να μπορέσουν να το σταματήσουν και να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Να ξέρουν τι γίνεται δηλαδή ώστε να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Έχετε επερώτηση? Όχι, ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τερέρο Σαλό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Γεωργέβα. Στην περίπτωση σοβαρών οικονομικών κρίσεων, κυρίως μετά από θεομηνίες, χρειαζόμαστε σωστικά συνεργεία, υγειονομική βοήθεια, ή νερό, αλλά πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε αρχές ε, που να είναι ορατές. Χρειαζόμαστε σαφές, σαφείς οδηγίες και εντολές, κάποιον που να λαμβάνει τα ενία και τον προγραμματισμό και ευθύνη στην άσκηση του έργου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι μπορεί να διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να υποστηρίξει σε τέτοιου είδους κρίσεις την σωστή διακυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί κάποιος που θα παίξει ηγετικό ρόλο για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μπορούμε να συστήσουμε κάποια επιτελεία, κάποιες ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν επιτόπου για τη σωστή διαχείριση των κρίσεων. Έχετε το λόγο κυρία υποψήφια Επίτροπε. Uh, uh, Συμφωνώ και χρειάζεται οπωσδήποτε. Αυτό που ακούμε και το ακούω και από τους συναδέλφων μας με την Παγκόσμια Τράπεζα ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας για το πώς ε, σχηματίζει η κυβέρνηση και τη δυνατότητα που έχει για να αντιμετωπίσει τα, προβλήματα. Κοιτάξτε, ούτως ή όλως δεν ήταν καμία κυβέρνηση της προκοπής. Τώρα συνέρχεται. Και θα είναι βέβαια κρίσιμο το αν θα μπορέσει να σταθεί ή όχι. Ε, κάτι άλλο όμως που πρέπει να, να σκεφτούμε είναι πώς μπορούμε να ανοίξουμε ευκαιρίες για το, η δράση του, ιδιωτικού τομέα, γιατί και πάλι αν ε, βασιστούμε μόνο στον δημόσιο τομέα και στη διεθνή στήριξη, δεν πρόκειται να αποκαταστήσουμε την ΙΤ ε, εύκολα. Θα είναι σίγουρα πολύ πιο μακρά, μακρύς ο αγώνας αυτός. Ιδιαίτερα όταν κινηθούμε στην, μετα... στην ανοικοδόμηση, θα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ώστε οι επιχειρήσεις να επανέλθουν. Υπήρξε κάποια... Υπήρξαν κάποιε ενθαρρυντικέ κινήσει στην ΑΕΤ ω προ αυτό, ώστε να μην ε, εξαλειφθούν τέτοιε δυνατότητε. Γιατί με τη δουλειά θα έρθει και αξιοπρέπεια και οι δουλειέ, οι θέσει δημιουργούνται όταν ε, ε, προωθείται και ο ιδιωτικό τομέα. Και αυτό το λέω όχι γιατί υποτιμώ την ανάγκη για παρέμβαση του δημόσιου τομέα και για διεθνού διεθνούς όχι. Γιατί ούτω ή άλλω αυτό ήταν. Διακόπτη πρόεδρο. Simplemente subrayar que, eh, por Θα ήθελα να επισημάνω ότι φυσικά θέλουμε να υποστηρίξουμε επιτόπου τους γηγενείς, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, γιατί αυτοί έχουν οι αρμόδιες αρχές τους φέρουν την ευθύνη του πληθυσμού. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε, να, να τους αντικαταστήσουμε στο ρόλο τους, αλλά να τους συνεπικουρήσουμε ώστε να μπορέσουν να κατευθύνουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στην αντιμετώπιση μιας κρίσης. Αυτό είναι το, η κατάλληλη στιγμή. Όταν οι θεσμικές δυνατότητες είναι πολύ χαλαρές. Χωρίς τέτοια στήριξη η χώρα δεν θα μπορούσε καν να σταθεί. Ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια της, αλλά θα ήταν ακόμα δυσκολότερο, ναι. Euh, Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν που συμμετέχει στη δική μας ε, ακρόαση συνδεδεμένα και την αντιπροσωπεύει η κυρία Αντίτα Στρέλα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζεωρζίεβα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των φυσικών καταστροφών στο ευρωπαϊκό έδαφος και στην ανακοίνωσή σας για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών που, ή των ανθρωπογενών καταστροφών η Κομισιόν επιβεβαιώνει πως θα διερευνηθεί δυνατότητα ανάπτυξης μιας ειδικής ε, πρωτοβουλίας για τις δασικές πυρκαγιές. Σημαίνει αυτό πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια οδηγία για τις δασικές πυρκαγιές όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμα του 2006 και θα είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που ήδη υπάρχει για τις πλημμύρες. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να απαντήσετε. Γίνεται πολλή δουλειά στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, από ό,τι κατάλαβα. Από την άποψη την αναπτυξιακή και από την άποψη της γεωργίας. Δεν ξέρω πόσο προοδευμένη είναι και δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Σίγουρα όταν δούμε τις πλημμύρες και δούμε αυτά τα πολύ ε, τα, τα φαινόμενα τόσο μεγάλων διαστάσεων και προσπαθήσεις να φτιάξεις μια οδηγία για να βοηθήσεις την ε, Ένωση να ανταποκριθεί. Ναι, αλλά αυτή είναι η ευκαιρία μου να είμαι σύντομη. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα ναι ή όχι σήμερα. Ε, αλλά θα επανέλθω, σας το υπόσχομαι. Έχετε το λόγο για επερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ήθελα επίσης να ξέρω, ήταν μια άλλη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το παρατηρητήριο για την ξηρασία, την απερίμωση και για τις πλημμύρες. Πιστεύετε πως ε, είναι σημαντική η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τις φυσικές θεομηνίες και πιο συγκεκριμένα να μπορέσουμε να ενεργήσουμε προλαμβάνοντας και όχι αντιδρώντας σε αυτές τις καταστροφές. Η κυρία Υποψήφια, Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ναι, φυσικά το να μπορούμε να προβλέψουμε ε, ε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πού υπάρχουν, πώς υπάρχουν και τι ε, θα μπορούσε να προσφέρει ένα τέτοιο κέντρο. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, όσο καλύτερη ενημέρωση έχουμε, τόσο πιθανότερο είναι να είμαστε έτοιμοι και να ανταποκριθούμε καταλήλως και θα μας κοστίσει και λιγότερο τόσο σε ανθρώπινο κόστος όσο και σε οικονομικό κόστος. Φτάνουμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι Catch the Eye, ερωτήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο θέμα της εσμίκρινσης, ε, της ανησυχητικής εσμίκρινσης ε, του ανθρωπιστικού τομέα και της παραβίασης, ε, της αυξανόμενης μάλλον παραβατικότητας όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο κύριος Μίτσελ Ελκ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η επιρροή του, ποινικού, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε σχέση, για παράδειγμα, με επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που σαφώς καταχρώνται και που ε, καταδικάζονται από το δικαστήριο αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί η συνεργασία. Φοβούμαι πως ε, εδώ μπαίνουμε σε ένα τομέα από την άποψη της ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω της αρχή τη ουδετερότητα και σκέφτομαι το Σουδάν, την απόπειρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να επιβάλλει την απόφασή του εκεί και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολε συνθήκες και είναι πολιτικό το ζήτημα, αλλά δεν είναι τμήμα του χαρτοφυλακίου αυτού. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι η κυρία Άστον θα ήταν ε, το σωστότερο άτομο στο οποίο να υποβάλλεται την ερώτηση αυτή. Δεν προσπαθώ να, το ξεφύγω, να ξεφύγω από την ερώτησή σας, αλλά νομίζω δεν εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιό μου. Κύριος Γεραίρος Σαλώμα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η προάσπιση του ανθρωπιστικού τομέα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια που θα γίνει στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Διά, ε, Όπως συζητήσαμε προηγουμένως, πραγματοποιείται αυτή η αναθεώρηση και θα δώσει τη δυνατότητα να ε, ανοιχτευτούν οι τονίες οι οποίο θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και να λάβει η χώρα ε, συμπληρωματική δράση ή επιτυχημένη δράση. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο ερώτημα είναι το πιο δύσκολο. Είναι το θέμα του συσχετισμού στρατηγικής και πολιτικής βοήθειας. η, η Ισπανική Προεδρία σκοπεύει να συζητήσει το θέμα αυτό και αν επιτύχει η πρόοδο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο η πρόοδο αυτή. Ο κ. Γεράς έχει το λόγο. Θα ήθελα να υποβάλλω την εξή ερώτηση, κυρία υποψήφια επίτροπε. Πριν από μερικέ χώρε το Μιανμάρ αρνήθηκε την πρόσβαση των ε, ε, εκπροσώπων ανθρωπιστικής βοήθεια μετά από μια καταστροφή. Καταλαβαίνω ότι είστε πάρα πολύ επιβλεκτικοί στην απάντηση. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε μία καταγραφή των απολυσθένων ζώων στην περίπτωση αυτή. Δεν ολοκληρώνω τη ρώτηση και διακόπτει ο πρόεδρος. Ναι, αυτό θα έξερα. Είναι κάτι που θα ξέρετε κατά περίπτωση. Θα πρέπει ανάλογα με το τι συμβαίνει να πάρουμε μία απόφαση σύμφωνα με το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Τότε η κρίση αυτή έγινε για κάποιους λόγους. Ο λόγος ήταν ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ υψηλά ε, ψηλές προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούν ε, αν πρόκειται να καλέσουμε στρατιωτική βοήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ενιαία λύση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε εκάστοτε τις ε, καταστάσεις και να σεβαστούμε τις αρχές βάσει των οποίων δημιουργούνται οι διεθνείς ανθρωπιστικές σχέσεις. Κύριο Στάς από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα εισαγωγικά σας σχόλια, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, είπατε ότι ε, θα πρέπει να πάρετε εκεί που η σχολική βία χρησιμοποιείται σαν ε, ένα όπλο στρατιωτικό. Αυτό γίνεται στο Ανατολικό Κονγκό κάθε μέρα. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Αυτή τη στιγμή τα μέτρα που έχουμε στα χέρια μας είναι να εξασφαλίσουμε όταν εμείς κάνουμε κάτι, δημιουργούμε δηλαδή ένα στρατόπεδο παραδείγματο χάρη, έχουμε κατά νου να μην εκθέσουμε τις γυναίκες σε κίνδυνο, να μειώσουμε δηλαδή έτσι αυτή τη σεξουαλική βία. Όταν εμείς ε, έχουμε πλατφόρμες επικοινωνίας και ε, ασφάλειας, πάλι έχουμε κατά νου το θέμα των γυναικών. Και βέβαια ερχόμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη για να προασπίσουμε το θέμα της χωρίς περισσότερης προσοχής, πιο έντονα εκφρασμένες δηλαδή απόψεις από όλους τους ηγέτες του κόσμου για το θέμα αυτό. Το μόνο πρακτικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε εκείνοι που είναι επιτόπου να το έχουν πάντα κατά νου. Η κυρία Θεοχάρους. Do you have the intention to impose sanctions on those countries, authorities? Σκοπεύετε να επιβάλλετε κάποιες κυρώσει κυρώσεις σε εκείνους που αρνούνται την ε, μεταβίβαση της βοήθεια σε εκείνους που τη χρειάζονται. <coughs> Απάντηση. Δεν έχω ένα τέτοιο μέσο στα χέρια μου. Λόγω ακριβώς τη ιδιαιτερότητας ε, και ανεξαρτησίας που πρέπει να τηρήσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά όπως είδαμε σε ακραίες περιπτώσεις κατάχρησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δώσει εκεί αναπτυξιακή βοήθεια όταν υπάρχει έντονη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μεταβιβάσω τις πληροφορίες για να μπορεί να ληφθεί υπόψη στις πολιτικές αποφάσεις του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής. Περνάμε τώρα στο τέταρτο τμήμα. Ο κύριος Σόλτερανς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στην λειτουργική διάσταση που θα πρέπει να υπάρχει για την εμπνόψη των ανθρωπιστικών κρίσεων. Η υποψήφια επίτροπος έχει κατά νου μια κατανομή του βάρους, ένα burden sharing στο εσωτερικό της Ένωσης. θα καλέσετε όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή να συμβάλλουν για να κατανομεί αυτή η βοήθεια. Η υποψήφια επίτροπος έχει το λόγο. Είμαι οπωσδήποτε υπέρ της κατανομής του βάρους και διαβλέπω και να μπορώ να παίξω ένα ρόλο στην προάσπιση πιο ενεργού συμμετοχή των νέων κρατών μελών. Εγώ προέρχομαι από μια νέα κράτος μέλος και έχω την υποχρέωση οι πολίτες της χώρας μου να έχουν περισσότερε πληροφορίες. Ακόμα και αν εμείς βρισκόμαστε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, υπάρχει εδώ μια δέσμευση που έχουμε να λάβει. Ακόμα δεν έχω αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν ε, συνδέεται με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη συμμετοχή και τον κατανομή του βάρους. Ελπίζω να το μάθω γρήγορα και να ενημερωθώ και από την Επιτροπή Ανάπτυξη για το θέμα αυτό τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Έχετε μια συμπληρωματική ερώτηση κύριε Γκέρντς. Όχι. Ωραία. Η κυρία Σάμπερ Σαστραμ του ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, το πρωτάριο θα πω ότι είναι πολύ ευχάριστο να συζητεί κανένας μαζί σας και ελπίζω δεν θα είναι η τελευταία φορά. Στις γραπτές σας απαντήσεις ε, λέτε ότι η πρόταση για ένα ευρωπαϊκό εθελοντικό σώμα θα την υποβάλλετε ακόμα φέτος. Ξέρετε πότε? Και ποια, δεν ποια μορφή θα έχει αυτό ακριβώς. Και θα θέλατε κι εσείς ήδη το 2011 να υπάρχει αυτό το εθελοντικό σώμα. Ε, μείνετε σε αυτή την αισιόδοξη πρόταση, κατά τη γνώμη μου. Απάντηση. Ναι, πραγματικά είναι αισιόδοξη. Αλλά βέβαια το χροδιάκμι είναι σημαντικό για το 2011 είναι το έτος του εθελοντιστού. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το σώμα, είναι καλό να υπάρχει τώρα και είναι κάτι που αναφέρεται στη παράγραφο 214 συνδείξη Λισαβόνα. Υπάρχει λοιπόν και θα πρέπει να φροντίσουμε να πραγματοποιηθεί. Δύο πράγματα θα πρέπει να έχουμε το νου. Το ένα είναι ο προπολογισμό. Το άλλο είναι ο στόχο του σώματο. Προπολογισμό γιατί δεν μπορεί να είναι τμήμα από τον προπολογισμό τη ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί αυτό θα ήταν άδικο προ εκείνου που θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από εκεί. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια θα ήταν η μορφή αυτού του σώματος. Γιατί προφανώς δεν θέλουμε να πάρουμε θελοντές και να τους στείλουμε σε κατάσταση κρίσης στην οποία χρειάζεται πάρα πολύ συγκεκριμένη προετοιμασία. Αλλά μπορούμε να έχουμε κάτι όπως πούμε μηχανική χωρίς σύνορα. Να έχουμε δηλαδή κατά το δυνατόν πολλούς εθελοντές που να θέλουν να εργαστούν χωρίς ε, κίνδυνο για την ασφαλειά σου, συρμανικό κόστος κλπ. Ίσως είμαι υπερβολικά ε, αισιόδοξη, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο στη συνθήκη και έχουμε το έτος του εθελοντισμού που επίκειται, θα πρέπει να κάνουμε κάτι πραγματικά. Αλλά χρειάζομαι προεβολογισμό και σωστό σχεδιασμό. Δύο πράγματα. Έχετε την πραγματική ερώτηση. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα υπάρχουν και δύσκολε συζητήσει με τα κράτη-μέλη από αυτού. Κοιτάξτε, η σημαντική λέξη είναι εθελοντικό σώμα. Γιατί εθελοντικό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι όλες οι χώρες, δεν θα πρέπει να είναι όλοι ο καθένας. Εθελοντικά. Πρέπει βέβαια να υπάρχει κάποια κινητοποίηση, να υπάρχουν κάποια χρήματα και όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν. Όποια κράτη-μέλη θέλουν να συμμετάσχουν, μόνο να συμμετάσχουν. Θα ήταν πολύ περίεργο να έχουμε ένα υποχρεωτικό εθελοντικό σώμα. Ο κ. Κάσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γεωργίευα, ξέρετε ότι είναι δύσκολο να κρίνουμε εμεί τι ικανότητε ενό υποψηφίου. Εγώ κάθομαι εδώ σε όλο το απόγευμα και έχω εντυπωσιαστεί από τι γνώσει σα, τη δημιότητά σου, τι ε, θαυμάσιες ικανότητε ικανότητε και το καταπληκτικό παράδειγμα τη ε, συνέπεια τη ε, πολιτική σα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να, ρωτήσει, να υποβάλει ερώτηση γιατί πρέπει να περάσουμε στη θετική διαδικασία επικύρωσης για σας τώρα. There were consensus. <laughs> ναι, συνένεση πραγματική. Okay, um, I, follow on uh, on my my, my line. Now we have um, Madame Eleni Teokorak η κυρία Ελένη Θεοχάρου από το ΕΛΚ. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κασμάν, ωστόσο θα κάνω μια ερώτηση. Είμαι εναντίον κάθε είδου στρατιωτική παρέμβασης και να το θυμάστε, οι Αμερικανοί δεν θα φύγουν ποτέ από την ΑΕΤ. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω αν προτίθεστε να οργανώσετε μια ανθρωπιστική δύναμη ταχείας ανάπτυξης, μια οργανωμένη δύναμη η οποία να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, δεδομένου ότι η Ευρώπη πιάστηκε απροετοίμαστη και στον Νότιο Λίβανο και στην Γάζα και στο τσουνάμι της ε, Σιρλάνκα και της Σουμάτρα και στην Αϊτή τώρα. Δηλαδή πέρα από τον εθελοντισμό που σίγουρα πάντα έχει κινδύνους ο εθελοντισμός χρειάζεται να υπάρχει και μια δύναμη οργανωμένη που να μπορεί να επιτελεί αυτή τη δουλειά. Υποψήφια Πέτρεβος έχει το λόγο. Η, η ιδέα μιας ε, ομάδας γρήγορης ανάπτυξης ή ανθρωπιστικής βοήθειας που αναφέρεται στην έκθεση Μπαρνιέ ακριβώς κινείται προς την κατεύθυνση μία μονάδα που αποτελείται από κράτη-μέλη και όπου υπάρχουν κενά, να συμπληρώνουν τα κενά από, από την Κομισιόν, από την Ένωση δηλαδή, στο σύνολό τη. Και χρειάζεται... είναι να το πω αλλιώ. Κατ' αυτό έχει νόημα. Αλλά αν κάτι δεν είχε γίνει τόσα χρόνια, θα πρέπει να υπάρχουν λόγοι γιατί δεν έχει γίνει. Και προτού καταλάβω τους λόγους αυτούς θα ήταν ανεύθυνο να τοποθετηθώ εγώ προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Οπωσδήποτε θα δεσμευτώ έντονα στο θέμα αυτό. Θα εξετάσω ποιε είναι οι συζήτησεις που θα γίνουν στο Συμβούλιο στις 11. Θα πρέπει να δούμε το θέμα με τη Βαρόνη Άστον να αφορά τη σημασία αυτές οι συζητήσεις αμέσως να περάσουν σε ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο και θα επανέλθω σε εσά όταν είναι σαφές γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και τι πρέπει να συμβεί για να λάβει χώρα, θα επανέλθω σε εσά. Έχετε με την ερώτηση. Μέχρι τότε προτίθεστε να εκδώσετε ένα τύπο διαβατηρίου ας πούμε για την προστασία όλων των εθελοντών οι οποίοι ε, πηγαίνουν με αρκετούς κινδύνους στις διάφορες χώρες και να διευκολύνεται το πέρασμα του στα δύσκολα σημεία, για παράδειγμα στο ΕΡΕΣ προ την Λόριδα τη Γάζα. Thank Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν είναι ένα θέμα για το οποίο έχω πληροφορίες. Ξέρω, στα Ηνωμένα Έθνη έχουμε ένα λεσέπασέ των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο σε ορισμένε χώρε είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουμε όσον αφορά τα έγγραφα που έχουν οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα. Όταν μάθω κάτι σχετικό, ευχαρίζω να επανέλθω και να σας πω τη γνώμη μου το λόγο κυρία Τόγια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε. Δώσατε σε όλους την εντύπωση ότι εκτός από τη διαχείριση των κρίσεων σας ενδιαφέρει και η φάση του προγραμματισμού και της προετοιμασίας. Είπατε να δώσουμε έμφαση στη δομή, να δούμε πώς ε, θα δραστηριοποιηθούμε, να διασφαλίσουμε πρόσφορες προϋποθέσεις. Αυτή την προσέγγιση την προληπτική ε, θέλω να θίξω και θέλω να θίξω ένα πρόβλημα. Υπάρχουν φυσικές ε, καταστροφές και ανθρωπογενείς ε, ε, καταστροφές ή λόγω της ε, ανάπτυξη. Πολλέ φορέ υπάρχουν, ε, τη υπανάπτυξη, μάλλον, υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν ε, ξηρασίες και ούτω καθεξής. Και έπειτα, μεγάλα σε περιοχές οι οποίες καλλιεργούνται εντατικά και μετά εγκαταλείπονται. Τι μπορούμε να κάνουμε, διακόπτη πρόεδρος. This, uh, this... Η ερώτηση αυτή ανάγεται στο σύνδεσμο που έχουν τα αίτια μιας καταστροφής και κάποιων επόμενων περιστάσεων που μπορείτε να διορθώσει τα, την καταστροφή ή να την επιδεινώσει. Εγώ, με βάση τις αρμοδιότητες μου, θα συνεργαστώ με τον Αρμόδιο Επιτροπό Ανάπτυξης, ώστε να επεξεργαστούμε τις αναπτυξιακές μας στρατηγικές υπό αυτό το πρίσμα, υπό το πρίσμα δηλαδή των συνεπειών που θα έχουν τέτοιε δράσει ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αηφορία, τον αντίκτυπο που θα έχουν οι δράσεις στους ανθρώπους, στους μετανάστες, στο βιωτικό επίπεδο και το θέμα της διαχείρισης, ε, τον κίνδυνο κρίσης. Αλλά δεν είναι αποκλειστική δική μου αρμοδιότητα θα συνεργαστώ με τον Αρμόδιο Επίτροπο και στις συζητήσεις που θα έχουμε και στο Σώμα των Επιτρόπων, ιδιαίτερα στη συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης, θα έχουμε αυτό το θέμα ως προτεραιότητά μας. Έχετε περώτηση κυρία Τόγια. Εγώ σας καλώ να ξεπερνάτε τις αυστηρές σας ε, ε, αρμοδιότητες, τουλάχιστον στο πλαίσιο της συνεργασίας και ε, του συντονισμού. Γιατί αν έχετε κάτι να πείτε, έξυπνο να το πείτε και να το κάνετε. Ε, και δηλαδή τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα πιο εύκολο είναι να μιλήσουμε, αλλά πιο δύσκολο είναι να διατηρήσουμε αυτά τα δικαιώματα σε περιπτώσεις ε, πήγουσας ανάγκης, βιασύνης κτλ. Just to be very clear. Ας είμαστε σαφείς. Εγώ εστιάζομαι σε αυτό το θέμα του καταμερισμού και του διαχωρισμού των ευθυνών, γιατί δεν θέλω να μου πει κανείς ότι το χαρτοφυλάκι της ανθρωπιστικής βοήθειας θα χρηματοδοτήσει η, την διαχείριση ύδατος στην Αφρική, γιατί έτσι θα απομυζήσει πόρους από το δικό μας στόχο για να χρηματοδοτήσει άλλους στόχους. Φυσικά θα δώσω έμφαση και στην ανάπτυξη όσο μπορώ ιδιαίτερα σε θέματα ανάπτυξη που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφές ή να επιτείνουν τις συνέπειες μιας καταστροφής. Ο κύριος Κριστιαν Πρέντα από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, έχω μία ερώτηση για τη συμπληρωματικότητα της ανθρωπιστικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ποια είναι η γνώμη σας σε ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, Υπάρχει συνοχή των δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεύτερον, ποια κατά τη γνώμη σας είναι η προστιθέμενη αξία που επιφέρει η ευρωπαϊκή δράση, η ευρωπαϊκή ένεση. Ενώση. Αυτά. Η υποψήφια επιτροπός. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βελτίωση στο θέμα της ε, παροχής ε, βοήθειας, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία της Άκρα. Είχαμε την διακήρυξη του Παρισιού μετά τη Συμφωνία της Άκρα και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τις διάφορες απαιτήσεις και τα κριτήρια και να δούμε ποιοι είναι οι εταίροι μας στον αναπτυξιακό κόσμο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία δίνουμε έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και στο τι προσφέρουν ε, οι δωρητές ή οι υπόλοιποι εταίροι. Πάντως ανέκαθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, ο σημαντικότερος δωρητής ό,τι αφορά την παρουσία της στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και με την ισχυρή αυτή παρουσία της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει σημαντική επιρροή. Ακόμη Έχει πειράσει ακόμη και την Παγκόσμια Τράπεζα ως προς τις δράσεις της. Τώρα που έγκυται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο τι έγκυται και το έχω δει και στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη προσοχή στο θέμα της ε, ποικιλομορφίας, ε, της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης, σε θέματα όπως γυναίκες και ανάπτυξη, σε υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ή σε προγράμματα μικρής εμβέλειας. Βέβαια, είναι σημαντικό να υπάρχει ένας τίτλος, μια ονομασία, ένας χαρακτηρισμός, γιατί τότε μπορούμε, όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση. Για θέματα περιβάλλοντος. Κανείς άλλος δεν έκανε τόσο σημαντικά πράγματα ώστε να προωθήσει το περιβάλλον και να το συμπεριλάβει στην αναπτυξιακή ατζέντα. Αλλά φυσικά για το περιβάλλον τίποτα δεν είναι αρκετό. Πάντως, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πραγματικά μεγάλο συγκριτικό πλονέκτημα για την ανάπτυξη. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Συγχαρητήρια θερμά κύριε Επίτροπε. We, we the um, participating... Τώρα έχουμε ερωτήσεις από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Την ερώτηση θα θέσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, ο κύριος Δομινίκ Μπόντις. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, απαντήσατε προηγουμένως σε μία ερώτηση για τη Λωρίδα της Γάζας. Σημείωσα την απάντηση, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί δυστυχώς η τραγωδία αυτή κρατάει πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί. Η Αίγυπτος, όπως ξέρετε, αποφάσισε να κλείσει την υπόγεια σύραγγα προς τη Λωρίδα της Γάζας, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούν σε απόλυτη απομόνωση. Γιατί δεν υπάρχει ανεφοδιασμός από το Ισραήλ, δεν, θα μπορεί να περάσει καν από το υπόγειο τούνελ της Αιγύπτου. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση έλλειψη ανεφοδιασμού, τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να δράσετε κάτι επιγόντως, γιατί αυτή η λανθάνουσα ανθρωπιστική κρίση που διαρκεί εδώ και πολύ καιρό θα πρέπει, ε, θα πρέπει να αποτρέψουμε στο να μετατραπεί σε μια νέα καταστροφή. Δύο λεπτά κύριε Επίτροπε για την απάντηση. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πολλά και περίπλοκα θέματα για τα οποία ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας δεν μπορεί να δράσει μόνος του, αλλά σε συνεργασία με το Σώμα των Επιτρόπων και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δεν πρόκειται να σας υποβάλω σήμερα συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο και απέναντι στους συναδέλφους με τους οποίους θα εξετάσω το θέμα πολύ πιο διεξοδικά. Από ανθρωπιστική άποψη πάντως υπάρχει ένα θέμα, το θέμα της πρόσβασης. Και αν δεν εξασφαλίσουμε και αν δεν ενισχύσουμε την πρόσβαση, τότε θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα και θα επιτείνουμε την εξαθλίωση αυτού του κόσμου. Αντιλαμβάνομαι το, το πρόβλημα και φυσικά θα υψώσω και εγώ τη φωνή μου, αλλά δεν θα πρέπει να είμαι μόνη μου. Δεν μπορώ μόνη μου να επιλύσω αυτό το ζήτημα που κρατάει εδώ και δεκαετίες. Και είναι θέμα ουσιαστικά εμπιστοσύνης μεταξύ δύο λαών. Πάντως θα εξασφαλίσω την προβολή αυτού του θέματος. Θα το υποβάλω σημαντική προτεραιότητα, ιδιαίτερα όταν το συζητήσω με τους ε, αρμόδιους επιτρόπους για τις εξωτερικές σχέσεις. Κύριε Μποντή, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Πριν από λίγο είπατε ότι σε κατεπίγουσες περιστάσεις, σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφύγει σε ορισμένα νομικά εργαλεία με βάση συμφωνίες σύνδεσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες ε, χώρες. Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πίεση προς, τη, προς το Ισραήλ, για παράδειγμα, για να ελαφρυνθεί η πίεση προς τη Γάζα και να εξασφαλιστεί αυτή η πρόσβαση που αναφέρατε προηγουμένως. Εγώ παρακολούθησα την κατάσταση ως ε, απλός πολίτης. Έξωθεν. Ε, και το θέμα φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω την αίσθηση πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δράση της και στη θέση που έλαβε ήταν ανέκαθε συνεπής. Και παρόλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε παρόλα αυτά να έχουμε κάποια επίδραση. Δεν είναι ότι έχουμε μείνει αμέτωχοι στην κατάσταση αυτή, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι μέσα χρησιμοποίησαμε. Αυτό το ζήτημα για μένα είναι πρωτόγνωρο. Και θα συζητήσω το θέμα ιδιαίτερα με τη Βαρόνια Άστον, που είναι αρμόδια για τα εξωτερικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μηχανισμοί ευρωπαϊκοί που θα μπορούσαμε να τους είχαμε χρησιμοποιήσει και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτά όλα θα τα ρωτήσω κυρίως από την κυρία Άστον και θα σας απαντήσω εν ευθέτω χρόνο. Υπάρχει επερώτηση τώρα. Με βάση ερωτήσει που έδωσαν οι πολιτικές ομάδες. Επαναλαμβάνω, ο χρόνος για τι απαντήσει είναι 1,5 λεπτό. Πρώτη ερώτηση. Κάποιες χώρες εκβιάζουν τη διεθνή κοινότητα και επίτηδες οδηγούν σε λιμοκτονία το λαό τους προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιήσουν τους δικούς σπόρους, όπως η Αιθιοπία. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Έχετε 1,5 λεπτό, κυρία Γεωργίευα, για να απαντήσετε στη δύσκολη αυτή ερώτηση. Όντως είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί άπτεται ενός βαθύτατου ηθικού διλήμματος. Ξέρουμε ότι η ίδια κυβέρνηση καταχράτα τους πολίτες τη και δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Και σίγουρα αυτοί που υπόκειται αυτή την καταπίεση υποφέρουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται τη βοήθεια. Όχι την κυβέρνηση δηλαδή, αλλά το λαό. Και να εκθέσουμε τις κυβερνήσεις, να τις θηλητεύσουμε, να τις εκθέσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι ότι θα μας ακούσουν άμεσα, αλλά έχουμε στα χέρια μας ως διεθνής κοινότητα ένα πολύ ισχυρό όργανο. Αν κάποιος ε, καταστρατηγεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο γίνεται παρείας στο διεθνές προσκήνιο. Μερικές φορές βέβαια οι κυβερνήσεις διαφορούν, αλλά άλλες φορές αρχίζουν, αρχίζουν και θορυβούνται γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερη ερώτηση από τα κόμματα. Πώς θα εξασφαλίσετε την, την αυτονομία της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να μην χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής για τη διαχείριση των κρίσεων. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν οι, ελπίζω, συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση είπε να μην μείνουν ρευστά τα σύνορα μεταξύ της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας, διαχείριση των κρίσεων, ε, διεθνούς συνεργασίες κτλ. Και όντως, μερικές φορές ε, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι το πιο σημαντικό γιατί εξαρτάται η ζωή πολλών ανθρώπων από την παροχή αυτής της βοήθειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Οπότε, στο νέο χαρτοφυλάκι που θα αναλάβω, αν όλα πάνε καλά, θα κρατήσω διαχωρισμένους στους δύο προϋπολογισμούς. Και υπάρχει και ένα νέο εργαλείο για την πολιτική προστασία που θα πρέπει να διαχωρίζεται από τον προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τι δυνατότητες υπάρχουν για να αξιοποιηθούν καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύετε ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το πιο σημαντικό είναι να συνεργαστώ με τον Αρμόδιο Επίτροπο Ανάπτυξης και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για την ανθρωπιστική ενίσχυση. Και χρειαζόμαστε πόρους και για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την ανάπτυξη. Αλλά πρώτα πρέπει να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και φυσικά με ενδιαφέρει η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς τις ανάγκες μας. Αν στα 9-10 χρόνια πρέπει να προσφύγουμε στα, αποθέματα, στα αποθεματικά μας για να χρηματοδοτήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, σημαίνει ότι δυστυχώ οι θεομηνίες είναι πιο συχνές και πιο οξύς από ό,τι στο παρελθόν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς θα το λάβουμε υπόψη. Σίγουρα υπάρχει συναγωνισμός ό,τι αφορά τους πόρους και προέρχομαι από μια παράδοση δημοσιονομικού συντηρητισμού και είμαι υπέρ της πολύ υπεύθυνη και ορθολογικής χρήσης των κονδυλίων. Αν τριπλασιαστούν όμως οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές και αν οι πόλεμοι εξακολουθήσουν είναι τόσο πολύ όσο στο παρελθόν, σημαίνει ότι οι ανάγκες μας θα επιταθούν και εξαιτία τη δημογραφικής ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι στι επόμενε δύο δεκαετίε ο παγκόσμιο πληθυσμό θα αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια και οι περισσότεροι θα διαβιούν στι αναπτυσσόμενε χώρε ή στις υπανάπτυκτε χώρε. Και θα εξακολουθούν οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται σε χαοτική κατάσταση, να ε, πλήττονται από θεομηνίε. Αν αυτή είναι όντω η τάση, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ταυτόχρονα πιστεύω στην καινοτομία, στην δημιουργικότητα στην εξασφάλιση χρηματοδότησης με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Δυστυχώς το παράδειγμα που θέλετε να μας δώσετε δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Τέλειωσε ο χρόνος. Ναι, ερώτηση. Μπορείτε να επεκταθείτε για το ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο ρόλος σας στη διεθνή συνεργασία και πώς αυτό θα συνοδεύεται, μάλλον θα συνδυαστεί με την εργασία του κ. Πίμπαλξ και της κυρίας Άστον των δύο άλλων επιτρόπων έχω κι άλλη μια παρόμοια ερώτηση. Το Κοινοβούλιο συχνά επικρίνεται ότι ε, ασχολείται υπερβολικά με τις δικές του αρμοδιότητες. Δεδομένου ότι πρώτα η Βαρόνη Άστον και έπειτα ο Επίτροπος Ντικούχτ μετέβησαν στην ΑΕΤ και τη σύγχυση που ε, κράτησε μετά. Εσείς είστε σαφείς για το ποιο κάνει τι στην Κομισιόν. Είστε σε θέση να έχετε πλήρη ευθύνη για τα ανθρωπιστικά ζητήματα ή θα αναθέσετε διάφορα θέματα στην, ε, ή μάλλον αντικαθιστάτε την κυρία Άστον. Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ είμαι επίτροπος ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτό και φυσικά όπως συζητήσαμε και σήμερα υπάρχουν πολλοί τομείς όπου θα βασιστώ στην Βαρόνια Άστον ώστε να διαβιβάσει τα μηνύματα, να λειτουργήσει ως αντιχείο για τη, τα θέματα τα δικά μου στους Υπουργούς Αμήνης και στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης. Αυτό θα το κάνω. Αλλά η ευθύνη μου, η ευθύνη μου ως ε, Επιτρόπου υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων θα είναι η, η δική μου ευθύνη. Θέλω επίσης να σας επαναλάβω κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά για τη διεθνή συνεργασία από τη στιγμή που σχετίζεται με τις κύριες, κύριες με ευθύνε και χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με αυτές τις ευθύνε, θα υπάρχει διεθνή συνεργασία. Αν θεωρηθεί πως δεν είμαι ανεξάρτητη και πως δεν είμαι ουδέτερη, δεν θα χρησιμεύσω στους ε, ε, εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα, αλλά ταυτόχρονα να δώσω στο σύνολο των επιτρόπων και εδώ στο Κοινοβούλιο ε, για θέματα τα οποία σχετίζονται με τις δικές μου ευθύνε, να τα προσφέρω ό,τι μπορώ να κάνω και μετά βεβαίως και να ε, τα προωθήσω στο διεθνή συνεργασία. Οι μελλοντικοί πρώην συναδελφοί μου της Παγκόσμιας Τράπεζας μου λένε ήδη ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ε, πρόγραμμα για τα ευάλωτα κράτη, για τα ευαίσθητα, εύθραυστα κράτη και λένε αν πας, αν πας θα συνεργαστείς μαζί μας ε, και είχα ήδη επαφές με διάφορους ε, διμερείς εταίρους. Δηλαδή, μπορούμε να, κατα... να φτιάξουμε ε, τομείς διεθνού συνεργασίας για τα διάφορα ζητήματα και κυρίως να το επεκτείνουμε και με τις περιφερειακή συνεργασία. Δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω με τη Ρωσία, αλλά μπορούμε να φτάσουμε στους νέους δότες, δωρητές. Αλλά δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Και τώρα περνάμε στον πέμπτο γύρο ερωταπαντήσεων. Και το λόγο έχει ο κύριος Νόρμπερντ Νάισερ από το Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στο στρατιωτικό και στο πολιτικό τομέα και να αναφερθώ συγκεκριμένα στο Αφγανιστάν. Το Γιάνναρη είχαμε τη διάσκεψη στο Λονδίνο στην οποία καθορίστηκε μια νέα στρατηγική και αναφέρθηκε συγκεκριμένα το θέμα της ενδυναμωμένης ε, ε, πολιτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν για την προώθηση της διαδικασίας συμφιλίωσης στο Αφγανιστάν. Ε, η επικοδόμηση αυτή και η ανθρωπιστική βοήθεια δίνονται κυρίως από την Ηνωμένα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αναρωτιέμαι κατά πόσο στον σύντονο χρόνο που είχατε, μια που είστε τόσο δραστήρια, Είχατε την εντύπωση να συλλέξετε κάποιες ιδέες για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Η υποψήφια προ... επίτροπος έχει το λόγο. There are some issues that are fairly clear. Υπάρχουν μερικά ζητήματα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, δεν είναι αποδεκτό για το, αποδεκτό για το στρατιωτικό σκέλος να δίνει ανθρωπιστική βοήθεια με τρόπο που προφανώς να μπερδεύει τα σύνορα, να συγχαίρει τα σύνορα ανάμεσα στην ε, στρατιωτική και την ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή, να λέμε ότι ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο, άμα είναι βαμμένο άσπρο, δεν θα βομβαρδιστεί. Από την άλλη πλευρά, όταν η εργαζόμενοι τη ανθρωπιστικής βοήθεια, ζητούν τη στρατιωτική στήριξη, ναι, τότε θα πρέπει να το σκεφτούμε και θα πρέπει να δοθούν και οι απαραίτητοι πόροι. Και, τότε, και μετά έχουμε όλο το σύμπαν που βρίσκεται ανάμεσα, όπου μια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε σχέση με το σε ποιο βαθμό θα δώσουμε ε, στρατιωτική βοήθεια ή στρατιωτική να μπουν στην ανθρωπιστική, στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Αν οι στρατιώτες του Αφγανιστάν έχουν μια ευκαιρία να χτίσουν ένα σχολείο, θα ήθελαν να το χτίσουν. Και θα ήταν και πιθανότατα πολύ καλό για τα παιδιά εκεί. Όμως μετά, Από την πλευρά της, ανα, της αναπτυξιακής βοήθειας έρχεται μια ομάδα που προσφέρει βοήθεια για να κατασκευάσει ένα σχολείο. Είναι αυτό ουδέτερο και ανεξάρτητο. Αυτό λέω, αυτό εννοούσα όταν μιλούσα για την Ισπανική Προεδρία και την συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να μείνει στον επίκεντρο της συζήτησης και θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια πορίσματα. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, μάλιστα. Στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες συζητούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θέλουν μία σαφή κατανομή μεταξύ της στρατιωγικής παρέμβασης ας πούμε και των πολιτικών στόχων και να μην υπάρχει καμία ανάμειξη μεταξύ των δύο αυτών. Εσείς πώς θα τον αντιμετωπίσετε. Επίτροπος. Ακριβώς αυτό είναι που εννοώ και εγώ. Ότι δηλαδή μπορεί να φαίνεται ότι είναι καλό, αλλά θέτει τον κόσμο σε κίνδυνο. Δηλαδή, οι στρατιώτες που βοηθούν ε, στην ανθρωπιστική πλευρά, καλό και ωραίο, αλλά οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια κινδυνεύουν έτσι. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις και να ληφθούν αποφάσεις για την ενδιάμεση αυτή φαιά περιοχή. Εμείς ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κάνει το στρατιωτικό σχέλος, να μην χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική πλατφόρμα για στρατιωτικές επιχειρήσεις και ναι, όταν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι χρειάζονται στήριξη, οι στρατιωτικοί να την έχουν. Η κυρία Στρίφλερ του ΕΛΚ. Εγώ θέλω να επανέλθω στην υπόθεση αυτών των παιδιών και των γυναικών στο Κογκό που βιάζονται καθημερινά. Και φυσικά πρέπει να γίνει απαραίτητο σε μια προληπτική δουλειά. Δεν πιστεύετε όμως πως αυτά τα εγκλήματα ενθαρρύνονται από την ατιμορρησία από πλευρά της κυβέρνησης, γιατί οι βιασμοί δεν γίνονται μόνο από τους στρατιωτικούς αλλά και από, από, από τους πολίτες. Δηλαδή, ε, πρόληψη θα υπάρξει στη βαθμό που παραμένει ε, μάλλον η αποτροπή θα είναι επαρκής από τη στιγμή που παραμένουν ατιμόρυτοι οι δράστες. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι βεβαίως το να, το να σε διαδικασία λογοδοσίας να θεωρηθούν υπόλογοι όλοι οι δράστες. Ο στρατό είναι υπεύθυνο για το τι κάνει η στρατιωτικοί, αλλά και οι διεθνεί ε, οργανώσει, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι υπεύθυνη για το τι κάνουν οι δικοί τη εργαζόμενοι. Κυρία Στίφλερ, έχετε ερώτηση. Ναι. Επερώτηση, όχι. Ωραία. Το λόγο έχει η κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα μια ερώτηση για τη Γάζα, αλλά σας έχει τεθεί πολλές φορές, ακόμα και να διατύπωνα διαφορετικά, δεν θα απαντούσατε με διαφορετικό τρόπο. Οπότε να σας θέσω μια άλλη ερώτηση. Εκτιμούμε πολύ την εμπειρία σας από την Παγκόσμια Τράπεζα και η ποιότητα των απαντήσεών σας ε, αποδεικνύει πως ήταν χρήσιμη για σας. Αλλά κάτι υπάρχει που το οποίο κάπως μας ε, ανησυχεί. Ανέκαθεν ήμασταν διστακτικοί στο Κοινοβούλιο σε σχέση με την, ε, χρήση των ε, ταμείων ε, γιατί πολλές φορές η ορατότητα της βοήθειας αυτής εξαφανίζεται. Εσείς ποια είναι η θέση σας για, αυτή για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον όσον αφορά την Παγκόσμια Τράπεζα, να σας πω ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ ορατοί από τα 24 μέλη του Συμβουλίου μας, του Διοικητικού Συμβουλίου μας, έχουμε ανάλογα με το χρόνο 8 ε, Ευρωπα... Ευρωπαίους μέλη και, και κάποιες φορές 9 μέλη. Πολύ ισχυρή φωνή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η Ευρώπη μάλιστα συνολικά είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος Τη Παγκόσμια Τράπεζα. και όταν συζητούσα με του συναδέλφου ότι θα έρθω στο Βρυξέλλε και τα λοιπά μου είπαν ότι η βασική συμφωνία είναι ότι τα γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας θα πρέπει να είναι στην πρωτεύουσα του βασικού μετόχου. Άρα έλεγα μάλλον θα με ακολουθήσετε κι εσείς. Ίσως χρειαστεί κι εσείς να με βοηθήσετε. Και καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι ναι, τα βάζετε όλα τα λεφτά μαζί, στο ίδιο καλάθι, αλλά δεν είναι τόσο ορατό. Το ίδιο σαν να έχει μια σημαία, ας πούμε, ένα γαλλικό project ή ένα ιταλικό project και ούτω καθεξής. Ε, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενημερώνει το κόσμο σε πού προέρχονται τα χρήματα. Για να σα ένα παράδειγμα, όταν δούλεψα στην Κίνα, με πήγαν σε ένα σχολείο το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα και Υποστηρίχθηκε και δεν θυμάμαι τότε από ποια χώρα, νομίζω από τη Γερμανία, διμερό. Στο σχολείο υπήρχε ένα μεγάλη, μια μεγάλη πλάκα που έλεγε Υποστηρίζεται και από την Παγκόσμια Τράπεζα και από την ε, Γερμανία. και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να αναγνωρίζονται τα project, αλλά δεν το κάνουμε. Και έχετε δίκιο ότι κάνουμε τι εκθέσει, δεν, δεν, δεν αναφέρουμε του πόρου, αλλά θα πρέπει, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει δημόσια στήριξη. Νικόπτη πρόέδρο. επερώτηση. <coughs> ναι, ίσως θα ξαναμιλήσω για την Γάζα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, όταν αναπτύχθηκε το τίμο με διάμεσο ε, μηχανισμό, η, προ... η Παγκόσμια Τράπεζα είχε το πρώτο ε, πτυχή, δηλαδή τα φάρμακα και την παιδεία, χρειάστηκε 1,5 χρόνο μέχρι ισότου να αναπτυχθούν αυτό το πρώτο ε, κομμάτι. Ενώ τα υπόλοιπα κομμάτια που τα είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ήδη αναπτυχθεί. Άρα χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Όντω. η Παγκόσμια Τράπεζα είναι πολύ συντηρητική για το πώς σχεδιάζει και εφαρμόζει τα project. Από τη μια πλευρά τα έχουμε πάει πολύ καλά και έχουμε χειριστεί την ε, διαφθορά. Ε, είμαι περήφανη για τα επιτεύγματα της τράπεζας, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνδυαστούν αυτά. Αυτό συμφωνώ. Ο κύριο Μάκελ Γκάλερ τώρα, του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι θέλετε να είσαστε πιο ενεργοί όσον αφορά τον τομέα της ε, ανθρωπιστική βοήθειας και τη αντιμετώπισης των κρίσεων. Ε, από τη δική σας εμπειρία μέχρι στιγμής ε, στη Διεθνή Τράπεζα, πού βλέπετε ελλείψη Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συνεργασία με διεθνείς ε, πολυμερείς οργανώσεις. Κατά τα άλλα, το βρίσκω λυπηρό που δεν θέλετε να απατήσετε τα χωράφια κανενός συναδέλφου του Άστον, του Πίπας, ε, του συναδέλφου για το περιβάλλον. Ε, γιατί εκείνη δεν είναι τόσο προσεκτική και τώρα το δικό σας χαρτοφυλάκο ε, λέγεται ε, διεθνή συνεργασία. Κρίμα είναι γιατί η Άστον ήταν χειρότερη από εσάς. Είσαστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν μην αφήσετε να σας πάρουν τις δικαιοδοσίες σας. Um, obviously I, I would take this Προφανώ ε, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το σχόλιο γιατί το τελευταίο που θα ήθελα να είμαι είναι να παραδώσω αυτά που κατά βάση ανήκουν στο δικό μου τομέα αρμοδιότητας. Γιατί στην περίπτωση δεν μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Γιατί αν είμαι, πρέπει να είμαι υπόλογη, πρέπει να είμαι και υπεύθυνη και θα πρέπει να έχω την ευκαιρία να κάνω τη δουλειά μου. Σας ευχαριστώ πάντως για την προειδοποίησή σας. Θα το λάβω σοβαρότατα υπόψη. Ευχαριστώ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, εκτός από τη διεθνή συνεργασία των κυβερνήσεων, εμείς ως βουλευτές έχουμε μια διεθνή κοινοβουλευτική διπλωματία μπορούμε να ελπίζουμε να σας δούμε συχνά εδώ στο κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε συνεργασία με τους συναδέλφους στην ε, ΑΚΕ, Ευρωμέτερ, ΛΑΤ, Ευρωνέστ και παραδείγματο χάρη θα μπορείτε τέλη Μαρτίου στην διάσκεψη ΑΚΕ στην Τενερίφα να σας καλέσουμε ήδη από τώρα που το κύριο θέμα συζήτησης είναι η ΑΕΤ. Η υποψήφια επίτροπος έχει το λόγο. Οπωσδήποτε θα είμαι παρούσα όπου χρειάζεται να είμαι παρούσα. Οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη πάρα πολύ σοβαρά το έργο μου. Και να πιστεύω πραγματικά ότι τα κοινοβούλια είναι η φωνή των πολιτών. Εδώ οι παρόντες έχουν εκλεγεί για το έργο τους αυτού. Πρέπει λοιπόν να είμαι υπόλογη σε εσά και θα πρέπει να συνεργαστώ επίσης και με τους εταίρους που έχουν ομολογώ ότι αυτό είναι ε, κάτι για το οποίο θα πρέπει να γνωρίσω καλύτερα. Να μάθω καλύτερα την αξία αυτών των σωμάτων και το τι μπορώ εγώ να προσφέρω. Αλλά πραγματικά θα αναλάβω την ευθύνη να είμαι παρούσα πολύ σοβαρά, όπου χρειάζεται. The last question is Mr. Gay Mitchell Τελευταία ερώτηση στον <laughs> κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ πρώτα. Σα υπέβαλα την πρώτη ερώτηση και έχω τη τιμή να σα υπέβαλα και την τελευταία ερώτηση. Εξ ονόματο των γνωστών τη ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών θα ήθελα να σα συγχαρώ για την παρουσίασή σα σήμερα. Σα εμπιστευόμαστε. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή πιστεύω μου δεν μπορούσε να καταρριφθεί το τείχος του Βερολίνου και όμως κατερρίφθη για να μπορέσουμε να κάνουμε ιστορία χρειαζόμαστε να μας εμπιστευτείτε κι εσείς. Εμείς εξ ονόματος των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι 30 που είμαστε εδώ, χρειαζόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας και χρειάζεται εσείς να συνεργαστείτε μαζί μας. Και εσείς και οι υπάλληλοι σας. Περιμένουμε να έχουμε δυνατότητα να σας ε, ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας, να συνεργαστούμε μαζί σας και έτσι θα μπορούμε πραγματικά πολλά να καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. We now have the Τώρα έχουμε τις συμπληρωματικές ερωτήσεις για τον τελευταίο αυτό γύρο των ερωτήσεων που θα σας διαβάσω. Νομίζω δεν, δεν υπήρχε <laughs> απάντηση, δεν χρειάζεται απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Μίτσο, δεν ήταν ερώτηση. Θα σας, υποβάλω, θα σας διαβάσω λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις των πολιτικών ομάδων. Ε, η νόμος της ε, ανθρωπιστικής ε, παρέμβασης έχει την ευθύνη να προστατευτεί η ε, ανθρωπιστική βοήθεια για να δώσει βοήθεια σε εκείνους που δεν έχουν φωνή και τι γίνεται όταν μια ε, λόγω χώρα αρνηθεί την πρόσβαση, πώς μπορείτε να ξεπεράσετε αυτή την άρνηση. Δύο λεπτά για την απάντηση σας παρακαλώ. Ε, με μεγάλη δυσκολία θα έπρεπε να απαντήσω, γιατί εν τελευταία αναλύση μόνο μια βιώσιμη ανάπτυξη η οποία δίνει στους πολίτες επιλογές, τους επιτρέπει να ευμερίσουν και οδηγεί σε δημοκρατικές κυβερνήσεις μόνο τότε δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα καταστροφών και ε, περιορισμό της πρόσβασης εκείνους που χρειάζονται τη βοήθεια περισσότερο. το δικό μου χαρτοφυλάκιο στην περίπτωση αυτή εξαρτάται στην επιτυχία των άλλων ε, πολιτικών της Ένωσης, ιδίως του χαρτοφυλακίου της ανάπτυξης και προτίθεμαι απόλυτα να υποστηρίξω τον Επίτροπο των Αρμόδιων για την Ανάπτυξη, γιατί μόνο εάν οι πολίτες έχουν η δυνατότητα επιλογής, είναι ελεύθερη, λειτουργεί η οικονομία τους, μόνο τότε μπορεί να τελειώσει αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ με βοηθάει η γραμματεία. Πολύ ευχαριστώ. Έχουμε το ολοκληρώσει αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις που υπέβαλαν, καθώς επίσης να ευχαριστήσω τον υποψήφια επίτροπο για τις απαντήσεις σας. Έχετε το λόγο κύριε Γεωργιέβα, εάν θέλετε να κάνετε κάποια ε, τελικά συμπεράσματα, πέντε λεπτά έχετε τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Πρόεδρε, ήταν πάρα πολύ πλούσια αυτή η συζήτηση δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλά να πω τώρα. Το μόνο που θα ήθελα να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε ε, να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε, να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες που παρουσιάσετε, που τις έχω καταγράψει εδώ. Μακρύς κατάλογος, αλλά οπωσδήποτε θα ε, εξετάσω περαιτέρω τις ιδέες και τις ερωτήσεις αυτές και μετά να διά Έχω τα πατήσει το χρόνο μου συχνά, τώρα θα είμαι σύντομη, αλλά θα ήθελα τελειώνοντας να σας ευχαριστήσω καταρχήν και να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Σήμερα, κατά σύμπτωση, είναι τα 81 ένατα γενέθλια της μητέρας μου. Uh, Κανονικά βέβαια θα έπρεπε να ήμουν κοντά τη σήμερα, αλλά τώρα είμαι εδώ και θα ήθελα να, κάνω, να σας κάνω μια υπόσχεση, μια υπόσχεση προς τη μητέρα μου. Μα η μητέρα μου πίστευε πάντα στην Ευρώπη. Έζησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τον κατακρισμό της Ευρώπης, αλλά πάντα πίστευε στην Ευρώπη και αυτό που ήθελε για μένα ήταν να μάθω γαλλικά, τα οποία δεν κατάφερα. Λοιπόν, η υπόσχεση που δίνει για τη μητέρα μου είναι εάν επιβεβαιωθεί η οικονομία θα προσπαθήσω να μάθω γαλλικά, στα γαλλικά η κυρία Γεωργίευα. Κύριε Αποψήφια Επίτροπε, είμαστε πάρα πολύ εδώ που θα θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μάθετε αυτή την πολύ ωραία γλώσσα. Πριν κλείσω τη συνεδρία, θα ήθελα να θυμίσω στους γνωστές ότι μια συνεδρίαση αξιολόγηση της ακρόσης θα γίνει σήμερα και κλεισμένο το θερόν στις 4.30 στην αίθουσα ASP 5G3. Πέρα στη συνεδρία σας. Καλό βράδυ.